Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Καλώς ήλθατε όλοι σας. Νομίζω ότι έχετε στα χέρια σας την ημερήσια διάταξη. Δεν ε, διατύπωσε κανένας ε, πρόθεση να γίνει κάποια τροποποίηση, επομένως μπορούμε να θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί για τις ανακοινώσεις για το δεύτερο σημείο. Θέλω να σας πω ότι μια μικρή αντιπροσωπεία μας πήγε στο Λονδίνο και μετά από κάποιες επισκέψεις είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Βουλή των Κοινοτήτων με μέλη τριών ε, επιτροπών από τη Βουλή των Λόρδων επίσης. Βρεθήκαμε και στην Τράπεζα της Αγγλίας και κάναμε και εκεί πέρα επαφές με τον, αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή, ε, ε, με τον, ε, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και μετά πήγαμε στο κτίριο της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρεθήκαμε σε επαφή με συνδικάτα και επίσης με τα μέσα ενημέρωσης στο τέλος. Όλα αυτά ήταν ενδιαφέρον διότι έγινε σαφές από αυτή την επίσκεψη ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του τραπεζοπιστωτικού συστήματος έχει κάθε ενδιαφέρον να αντιμετωπιστεί αυτή η χρηματοοικονομική κρίση η οποία έχει παρουσιαστεί στις εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωση ως ευρώ, κρίση του ευρώ να επιληθεί αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο παρά το γεγονό ότι δεν ανέκει στη ζώνη του ευρώ είναι φανερό ότι έχει κάθε ενδιαφέρον στο να παραμείνει σταθερή η ζώνη του ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, θα κάνουμε μια αντίστοιχη επαφή με την ε, γερμανική Bundestag στο Βερολίνο. Οι αρμόδιες επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα των οικονομικών θεμάτων μας είπαν ότι μόνο την ε, Τρίτη το μεσημέρι μπορούμε να συναντηθούμε μαζί τους και αιτήσει του Σέργιο Κομφεράτη κανονίσαμε να υπάρχει και διερμηνία αλλά θα υπάρχει διερμηνία μόνο γερμανικά-αγγλικά, αγγλικά-γερμανικά. Όποιος λοιπόν μπορεί να καλυφθεί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το αναφέρει στο Προεδρείο μας και θα κανονιστεί αυτό το ταξίδι. Είναι μια πολύ σύντομη επαφή ή είναι απλώς ένα γεύμα εργασίας ουσιαστικά. Επίσης για το Λονδίνο θέλω να σας αναφέρω που δεν είχα ποτέ συναντηθεί με εκπροσώπους της Βολής των Λόρδων ήταν όχι μονάχα παιδαγωγικό και ενδιαφέρον, αλλά και κάτι το οποίο με εντυπωσίασε και μου προξένησε ακόμα και έκπληξη, το πόσο δηλαδή συστηματικά, πόσο εντατικά τα μέλη των τριών αυτών επιτροπών της Βουλής των Λόρδων είχαν προετοιμάσει τις συζητήσεις μαζί μας. Εγώ είχα μελετήσει πολύ καλά την έκθεση της ε, Περβανος Μπερές. Αυτοί ξέρανε απ' έξω και ανακατοτά διάφορα άρθρα της ε, έκθεσης αυτής Οπότε ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι για να μας απαντήσουν στα ερωτήματα που τους θέσαμε. Και έρχομαι στα σημερινά μας. Έχουμε δύο σημεία τα οποία θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν το θέμα των ε, παγκοσμίων άνο, άνισομεριών και της παγκόσμιας μορφής συντονισμού και διακυβέρνησης. Και εδώ τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει σε σχέση με το υπάρχον σύστημα νομισματικών ισοτιμιών αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να τροποποιηθεί αυτό το σύστημα, αν υπάρχει μάλλον από χρόν λόγος για να τροποποιηθεί αυτό το σύστημα για να ξεπεραστούν αν όχι ολοκληρωτικά αλλά τουλάχιστον μερικά οι ανισομέρειες και να αποφευθούν κρίσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν από νομισματικές ανισομέρειες και έχουμε εδώ τον κύριο Μπέξ ο οποίος είναι διευθυντής αρμόδιος για διεθνείς ε, σχέσεις στα χρηματοοικονομικά θέματα και τον ε, παγκόσμιο συντονισμό σε χρηματοοικονομικό επίπεδο στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και θα λάβει το λόγο και για τα δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν τόσο τις παγκόσμιες ανισομέρειες όπως και το ζήτημα ενός νέου νομισματικού συστήματος με μια παρουσίαση περίπου 15 λεπτών. Μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως σας είπε και ο Πρόεδρός σας, νομίζω είναι λογικό να διαχωρίσουμε τη συζήτηση αυτών των δύο θεμάτων, παρότι είναι αλληλένδετα και θα διαπιστώσετε στις ομιλίες μου ότι θα χρειαστεί να κάνω παραπομπές στο άλλο θέμα θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη συζήτηση αυτών των δύο θεμάτων, αλλά και τα δύο διεξοδικά πρέπει να τα συζητήσουμε. Για τις παγκόσμιες ανισότητες, ανισομέρειες, στους, στις τρέχουσες συναλλαγές. Ε, εδώ και καιρό συζητούμε αυτό το θέμα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 άρχισαν να μας απασχολούν σε παγκόσμια επίπεδα. Τότε υπήρχαν μεγάλες ε, κεφαλαιακές ροές ε, προς το Ηνωμένο Βασίλειο, προς τη ΣΥΠΑ και δημιουργήθηκαν σοβαρά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών. Τώρα, στον αντίποδα, Κίνα και η Ιαπωνία αυτές μεγάλωσαν, ε, διεύναν τα πλεονάσματά τους ε, περαιτέρω. Όλη την περασμένη δεκαετία υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες σε αυτούς που εκπονούν την πολιτική, καθώς και στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν για τα ελλείμματα, αλλά φοβούμασταν ότι θα ήταν απότομες και θα οδηγούσαν σε ισχυρή υποτίμηση του δολαρίου και την απότομη αναστροφή των κεφαλαιακών ροών, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει ε, σε ύφεση, μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Παρατηρήθηκε η μεγάλη κάμψη της ανάπτυξης βέβαια, αλλά για διαφορετικούς λόγους, λόγω της παγκόσμιας δηλαδή χρηματοοικονομικής ε, κρίσης. Αυτά που διαπιστώσαμε τότε, το 2009, μας οδήγησαν στη διαπίστωση ότι όντως είχαν ε, διωγκωθεί τα ελλείμματα στις τρέχουσες συναλλαγές και είναι μειονέκτημα και πλεονέκτημα ταυτόχρονα. Τώρα εξερχονται οι χώρες από την ε, κρίση και ε, διωγγώνονται αυτές οι ανισομέρειες. Ε, δηλαδή οι τάσεις που υπήρχαν πριν από την κρίση αναφύονται και πάλι. Σε παγκόσμιο επίπεδο διαπιστούμε μεγάλες ανισότητες. Βλέπετε στον πίνακα, σε αυτό το, στο παράρτημα του εγγράφου που δώσαμε στην Επιτροπή σας, στον πίνακα λοιπόν Βλέπετε τα στοιχεία και θα ήθελα να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για την Κίνα. Φαίνεται ότι είναι υποέλεγχο η κατάσταση, 5% για τα επόμενα χρόνια το, είναι το έλλειμμα, αλλά στο μέλλον να ξέρετε ότι το Δήμο το έχει κάνει προβλέψεις για πολύ υψηλότερο έλλειμμα, 7-8% του ΑΕΠ. Δεύτερον, ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, ακόμη και αν ε, μιλάμε για το πλεόνασμα των τρεχουσών συναλλαγών που κυμαίνεται στο 5%, αυτό οδηγεί σε μεγάλη αύξηση σε ονομαστικές τιμές. Το ίδιο και για την αύξηση του ΑΕΠ. Αναμένεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ στην Κίνα τα επόμενα χρόνια. για να δούμε τώρα τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για το 2010 με τα στοιχεία που έχουμε ε, μηνιαίως για το διεθνές εμπόριο και βασισμένοι στις μελέτες ε, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι για το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια ανάπτυξη ότι επιβραδύνονται. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε οριακά προς τα πάνω ε, το προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη από 7% στο 7,1% ενώ ε, για το 2011 11 αναθεωρήθηκε επίση το ποσοστό για την παγκόσμια ανάπτυξη από 4,2 στα 4,7%. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της Επιτροπής μας, τις προβλέψεις που κάναμε το φθινόπερο. Παρ' όλα αυτά είναι επισφαλής η κατάσταση, ε, κυρίως για τις οικονομίες όπου είναι, παραμένει υψηλή ανεργία. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε τις αναδυόμενες ε, οικονομίες ε, που δείχνουν μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη κυρίως στην Ασία και στην Λατινική Αμερική, παρότι και εκεί επιβραδύνεται η ανα... Ε, επιβραδύνονται οι αναπτυξιακοί ρυθμοί. Στις περισσότερες οικονομίες ε, υπάρχει ισχυρός πληθωρισμός ε, στην Ασία είναι ισχυρότερε οι πληθωριστικέ πιέσει λόγω τη ε, τιμή των αγαθών, των τροφίμων και τη ενέργεια ε, που παραμένουν σε χαρακτηριστικά υψηλά επίπεδα λόγω τη ισχυρή ανάπτυξη. Στι παγκόσμιε αγορέ βελτιώθηκαν κάπω τα πράγματα του τελευταίου μήνε. Ε, παρότι υπάρχει μια νευρικότητα και είδαμε ε, κάποιες ε, εκδηλώσεις αυτής της νευρικότητας για να αποφευθούν κίνδυνοι σε σχέση με τα ασφάλιστρα κινδύνου. Τώρα θα ήθελα να σας πω για την οικονομική ανάκαμψη, παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, ότι παρουσιάζει ισχυρές ανισότητες και επίσης υπάρχουν και κίνδυνοι, παρότι γενικότερα είναι βίωνες οι προβλέψεις και οι προοπτικές. Πρώτον, ε, το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η αξία των βασικών αγαθών. Ε, η τιμή των βασικών αγαθών. Αυτός είναι και ο βασικός κίνδυνος παρά την ε, παγκόσμια ανάκαμψη. Σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες κυρίως παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, δηλαδή πιέζονται προς τα πάνω σχεδόν όλες ε, οι τιμές, είτε μιλάμε για τρόφιμα είτε για μέταλλα και λόγω αυτού ενισχύονται ήδη υψηλές τιμές και μπορεί να εκτροχιαστεί αυτή η επισφαλής οικονομική ανάπτυξη και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και να αποτελέσει κίνδυνο για την αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος ε, του αναπτυγμένου κόσμου. Τώρα επανέρχομαι στο αρχικό θέμα, το θέμα μας για σήμερα, η τιμή ε, των εμπορευμάτων αυξάνεται και έτσι αυξάνεται η πίεση προς τους εισαγωγείς και ε, οι εξαγωγικές χώρες φυσικά διευρύνουν έτσι, ε, περαιτέρω το πλεόνασμα των τραγουστών συναλλαγών. Κάτι άλλο τώρα, η αστάθεια που παρατηρείται στις κεφαλαιακές ε, ροές, πολλές αναδυόμενες οικονομίες συσσωρεύουν τα αποθεματικά τους σε ξένα νομίσματα και αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλες μεταβολές των ισοτιμιών και αυτό δεν αντικατοπτρίζει αν θέλετε τα βασικά οικονομικά μεγέθη μόνο. Σα είπα ότι υπάρχει σχέση με το επόμενο θέμα μας, δηλαδή το διεθνέ Νομισματικό Σύστημα, αλλά διεξοδικότερα θα ε, συζητήσουμε αυτό το θέμα αργότερα. Τρίτος κίνδυνο, ο κίνδυνο τη ε, δημοσιονομική εξυγίανση ε, σε πολλές σημαντικέ, ανεπτυγμένε οικονομίε, είπα κυρίω και η Ιαπωνία. Ε, τα τρέχοντα μεγάλα ελλείμματα, αν ε, εξακολουθήσουν να εφίστανται μακροπρόθεσμα, ε, τότε θα οδηγηθούν αυτές οι χώρες σε μεγάλα επίπεδα δημοσίου χρέους, κυρίως για την Ιαπωνία και αυτό πλήττει την ε, ε, αναπτυξιακή, αν θέλετε, ικανότητα αυτών των χωρών και δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση των δαπανών που σχετίζονται με την γύρανση του πληθυσμού, κυρίως στην Ιαπωνία. Ε, τώρα, διωγγώνονται αυτές οι ανισότητες αν δεν κάνουμε τίποτα και Γι' αυτό το λόγο ο βασικός κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία είναι η έλλειψη ε, διόρθωσης, η έλλειψη ρύθμισης αν θέλετε αυτών των ανισοτήτων που παρατηρούνται. Με τι θα έμοιαζαν οι λύσεις. Ε, πρώτον, εφόσον πρόκειται για αμυγός ε, παγκόσμιο πρόβλημα, η απάντηση, η λύση πρέπει να είναι παγκόσμια. Πολυμερής δράση, συνέργειες, η ομάδα G20 που αυτοανακηρύχθηκε σε βασικό φόρουμ για παγκόσμιο οικονομικό συντονισμό πρεσβεύει ότι είναι στην καλύτερη δυνατή θέση για να δώσει μία απάντηση. Εξάλλου είναι και το μόνο φόρουμ έτσι, που μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέρσι το G20 ε, συμφώνησε επί ενός σχεδίου δράση τεσσάρων σημείων ε, για την τόνωση της ε, οικονομικής ανάπτυξης και τη διόρθωση των οικονομικών ανισορροπιών. Καταρχά, θα πρέπει να υπάρξει εξυγίανση των δημοσιονομικών. Έγιναν δύο συναντήσεις κορυφή, όχι μόνο στη Σεούλα, αλλά ε, και τον Ιούνιο έγινε μια συνάντηση και υποτίθεται ότι ανέλαβαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την ε, κατά το ίμιση μείωση των ελλημάτων τους μέχρι το 2013 και τη μείωση επίσης διαδίου του ποσοστού του χρέους στο ΑΕΠ. Αυτό το οποίο βλέπουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι ότι δεν επιτυγχάνει τους στόχους της. Στο Τορόντο υπόθηκε επίσης ότι ορισμένες ευάλωτες χώρες και εννοείται ευρωπαϊκές θα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα στον τομέα της εξυγίανσης των δημοσιονομικών. Το δεύτερο στοιχείο του προγράμματος δράσης της ομάδας των 20 είναι να υπάρξουν πολιτικές για την υποστήριξη της κατανάλωσης σε χώρες αναδυόμενες με πλεόνασμα. Σε ορισμένες χώρες, και εδώ εννοούμε την Κίνα, σε ορισμένες χώρες θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στις, ε, στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου δηλαδή και επίσης ε, αύξηση των δαπανών για υποδομές. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι όλες οι χώρες της ομάδας των 20 θα πρέπει να υιοθετήσουν διαρθρωτικές αλλαγές για την αύξηση και στήριξη των προοπτικών ανάπτυξής τους ιδιαίτερα στην Ευρώπη, θα πρέπει να αυξήσουμε το δυναμικό αναπτυξιακό το οποίο έχουμε και ταυτόχρονα η ομάδα των 20 θα πρέπει να επιτελέσει πρόοδο στην αποκατάσταση της διεθνού ζήτησης. Ε, στα πλαίσια αυτά συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την αντιμετώπιση των διεθνών ανισορροπιών μέχρι ε, την επόμενη συνάντηση τον Νοέμβριο στις Κάνες του 2011. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή αυτού του προγράμματος δράσης με τέσσερα σημεία σημαίνει ότι δημιουργούμε καταρχάς αυτό το οποίο νομίζουμε ότι είναι μια συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτής της ανάπτυξης τώρα γιατί όλα αυτά τα στοιχεία θα συζητηθούν στις άλλες συναντήσεις τις οποίες οργανώνει η Επιτροπή σας ή σε συναντήσεις τις οποίες είχατε ήδη. Να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι αφορά τις διαφθορτικές αλλαγές, την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, το θέμα του πακέτου μεταρρύθμισης στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, της ενίσχυσης των μηχανισμών ασφαλείας και την ενίσχυση του διακανονιστικού και εποπτιακού σε εισαγωγικά πλαισίου. Προσπαθούμε λοιπόν και από δική μα πλευρά να ενισχύσουμε τι προσπάθειές μα και ελπίζουμε ότι οι άλλες χώρες θα κάνουν το ίδιο. Θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι ο βασικό συνεισφορέα στι ε, διεθνεί ελλείψεις ε, ισορροπιών δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίω η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί δηλαδή. Για την Κίνα θα πρέπει να ενισχύσει τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχει, θα πρέπει να προωθήσει την οικονομική απελευθέρωση στην αγορά της και θα πρέπει επίσης να εισαγάγει μέτρα με στόχο την μείωση ε, του φαινομένου της μη απόδοσης μερισμάτων όταν υπάρχουν κέρδη σε μια ε, εισηγμένη επιχείρηση. Συνεπώς λοιπόν, έτσι το ΡΕΝΜΙ, το νόμισμα της Κίνας θα μπορέσει να πάρει την σωστή του αξία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί θα πρέπει να διασφαλιστεί μια αποκατάσταση της ισορροπίας του αναπτυξιακού δυναμικού μέσω της αύξησης ε, της αποταμίευσης σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να εφαρμοστεί επίσης και ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσιονομικής αποκατάστασης και για την αύξηση των αποταμιεύσεων σε επίπεδο δημοσίου. Ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ενέργεια και το περιβάλλον υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν γιατί αν βελτιωθούν τα πράγματα εκεί θα οδηγηθούμε σε μια καλύτερη αηφορία θα έλεγα της ιδιωτικής, εισαγωγικά το αηφορία της ιδιωτικής κατανάλωσης στη συγκεκριμένη αυτή χώρα. Τώρα, τι γίνεται με άλλες χώρες ε, οι οποίες έχουν ε, πλεόνασμα. Η Ιαπωνία, σαν παράδειγμα. Και εκεί θα πρέπει να εισαχθούν μέτρα διαρθρωτικών αλλαγών για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. Θα πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ σημαντική πρόοδος και σε αλλαγές στην αγορά εργασίας έτσι ώστε οι πραγματικοί μισθοί στις χώρες αυτές να αυξάνονται ανάλογα με τα κέρδη της παραγωγικότητας. Και αυτό με τη σειρά του θα πρέπει να βοηθήσει στην ενίσχυση της ιδιωτικής <clears throat> μέσω πρόθεσμα. Παράλληλα, νομίζουμε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου χώρες θα πρέπει να κάνουν περισσότερες ε, προσπάθειες για να διαφοροποιήσουν τις πηγές ανάπτυξής τους. Ορισμένες χώρες θα πρέπει να αυξήσουν τις δαπάνες τους στον τομέα των υποδομών, άλλες στον τομέα της εκπαίδευσης, έτσι ώστε σε ένα ε, ε, μέσο πρόθεσμο μέλλον να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και τη μακροοικονομική τους σταθερότητα. Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, έχω ήδη μακρηγορήσει να πω λίγα λόγια για κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει ελπίζω. Μία λόγια δηλαδή για τη συνάντηση της ομάδας των 20 που είχαμε ε, στο Παρίσι στα μέσα Ιανουαρίου. Η πρώτη συνάντηση υπό τη Γαλλική Προεδρία σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε σχέση με τις λεγόμενες ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές αντιμετώπισης της έλλειψης ισορροπιών. Στο Παρίσι αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε δύο φάσεις. Σε μια πρώτη φάση οι χώρες οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται και θα πρέπει να υφίστανται ανάλυση σε βάθος τα οικονομικά τους και τα δημοσιονομικά τους θα πρέπει φυσικά πρώτα να γίνουν αντικείμενο επιλογής, να ανοιχτευθούν δηλαδή οι χώρες στις οποίες θα γίνει η μελέτη αυτή σε βάθος. δεύτερη φάση είναι μέσω αυτής της μελέτης σε βάθος να δούμε ποια είναι η αιτία αυτών των εξωτερικών ανισοτήτων και πώς μπορούμε να κάνουμε συστάσεις στις συγκεκριμένες χώρες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αιτίες βάθους θα έλεγα οι οποίες προκαλούν προβλήματα δυσδιαχείρισης των οικονομικών. Υπήρξαν αντιθέσεις από πλευράς Κίνας ιδιαίτερα, Ρωσίας επίσης, Τουρκίας για τα μέτρα τα οποία προτείναμε. Αλλά παρόλα αυτά η Προεδρία η Γαλλική κατάφερε να οδηγηθούμε σε αυτές τις συμβιβαστικές και ενδιαφέρουσες λύσεις. Αυτή η αντιμετώπιση του προβλήματος σε δύο φάσεις προτάθηκε πρώτον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σεούλ, στη συνάντηση της ομάδας των 20 και επηρεάζεται και από τις δικές μας περίπλοκες διαδικασίες υπερβολικών ε, πλεονασμάτων και ε, είναι κάτι το οποίο θα ανήκει και στο πακέτο μεταρρύθμισης των μεθόδων διακυβέρνησης οικονομικής που θα προτείνει συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας είναι μεν φιλόδοξο αλλά είναι εφικτό. Θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τις συστάσεις αυτές και σε επίπεδο ηγετών στη συνάντησή τους στις Κάνες τον μήνα Νοέμβριο του 2011, του ενεστώτος έτους Υπάρχει ένα πλαίσιο εργασία επίσης, μια ομάδα εργασίας συγγνώμη, ε, στο εσωτερικό της ομάδας των 20, του G20, το οποίο θα συνεργαστεί και με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για την κατάρτιση των δικτών που θα πρέπει να υιοθετηθούν έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή και να ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα από αυτή τη διαδικασία σε δύο βήματα την οποία προανέφερα. Όπω είπαμε, το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσουμε, να ανοιχνεύσουμε τι προβληματικέ χώρε και να ξεχωρίσουμε τι χώρε οι οποίε δεν έχουν πρόβλημα. Αφού συμφωνήσουμε στη συνάντηση που θα γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου για τα επίπεδα και τους δείκτες, τότε τον μήνα Απρίλιο όταν υπάρξει η συνάντηση Υπουργών Οικονομικών της ομάδας των 20 στη Washington θα, θα έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα και θα προχωρήσουμε με την ανάλυση μας. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι φιλόδοξο, αλλά δεν θα είναι εύκολο ή το να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, κυρίω γιατί υπάρχει μεγάλη διστακτικότητα, μεγάλη αντίσταση από την πλευρά τη Κίνα, που είναι ένα μεγάλο παίκτη. Χωρί την Κίνα δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό των παγκοσμίων ανισομεριών. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέξ, για την πλήρη αυτή παρουσίαση στο θέμα αυτό. Εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε με, τον, με την εισηγήτρια, την Περβάον ε, Μπερές, και μετά να ακολουθήσουμε μια σειρά μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Έχω τον κύριο Χέκμαρ, την Ελίζα Φερέρα και τον Όλι Σμιτ που θέλουν να λάβουν τον λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που έρχεται σε μια στιγμή που είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ό,τι αφορά και την Επιτροπή μας, όπου έχουμε ακριβώς και εμείς τις ίδιες ανησυχίες και συμμερίζομαι ιδιαίτερα αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τον χειμερικό χαρακτήρα της ε, πεποίθησης ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες και ανισομέρειες σοβούσης της κρίσης. Μέσα στα άλλα στοιχεία Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε όλες αυτές τις πτυχές. Η Κομισιόν έχει αναλύσει την κατάσταση του κρατικού χρέους σε διάφορες χώρες, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη και τον αντίκτυπο της κρίσης που ουσιαστικά επιδίνωσε τα πράγματα. Κάποιες φορές η κρίση μειώνει την πίεση που υπήρχε στα δημόσια οικονομικά, σε άλλες περιπτώσεις τα έκανε χειρότερα, ιδιαίτερα σε σχέση με το κρατικό χρέας. Αν δεχτούμε το στιγμίο χαρακτήρα ορισμένων καταστάσεων λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούμε και πιο ευρέως σε σχέση με το κρατικό χρέος. Όπως σας είπα, η Ευρώπη δεν ήταν από εκεί που ξεκίνησε η κρίση. Μετά την κρίση η Ευρώπη έκανε πολλές προσπάθειες για να τακτοποιήσει τα πράγματα στο εσωτερικό της και να πείσει και τους παγκόσμιους εταίρους της. Δυστυχώς όμως, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τον οδικό χάρτη που έχουμε εισαγάγει για τα θέματα αυτά φαίνεται ότι δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχουν καταρχήν κάποιες πολιτικές συμφωνίες για τις ε, πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τις προϋποθέσεις τους. Δεν είναι το θέμα που μας απασχολεί σήμερα και θα μπω σε λεπτομέρειες. Παραμένει όμως μία δυσκολία που είναι <clears throat> οι προϋποθέσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να λειτουργήσει κάτι σε πολυμερές επίπεδο. Εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφέρον να λειτουργήσουν οι πολυμερείς δομές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά ακόμα και αν κάνουμε εμεί τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, αν ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση, βελτιώσουμε τις εποπτικές μας δομές, ακόμα και τότε θα παραμείνει ένα πρόβλημα οργάνωσης, ε, εκδήλωσης προς τα έξω τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν έχουμε παρουσία στους G20, δεν έχουμε το ειδικό βάρος που θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί το πιο ουσιαστικό από τις συνόδους των G20 είναι ότι γίνεται μία, έγινε και μία συνέντευξη τύπου. Αλλά εκεί στη συνέντευξη τύπου για τα προβλήματα αυτά δεν ελέγχθη ούτε φωνή ούτε ακρόαση σε σχέση με το ευρώ. Το ευρώ εμάς μας υποχρεώνει να έχουμε κάποιο ρόλο μέσα στις, ε, στους 20 Για τους άλλους <clears throat> παγκόσμιους παίκτες τα πράγματα είναι αρκετά μπερδευμένα βέβαια. Και έχω και μερικές ανησυχίες σε σχέση με τους άλλους εταίρους μας. Έναντι των Αμερικανών. Εγώ εντυπωσιάστηκα που στην αρχή της κρίσης για λόγους εσωτερικής πολιτικής των Πολιτειών, που δεν θέλω να αρνηθώ την ύπαρξή τους γιατί στι ΗΠΑ η ανεργία έχει φτάσει σε επίπεδα δυσκόλως ανεκτά, γιατί το σύστημα ευμάριάς τους και κοινωνικών παροχών βασίζεται στην πλήρη απασχόληση. Το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης απασχόλησης είναι ότι δημιουργήσαν ένα σχέδιο ανάκαμψης με το οποίο έχουν οξύνει ακόμα περισσότερο την παγκόσμια ανισομέρεια. Αυτό δεν μπορούμε να το συζητήσουμε με τους Αμερικανούς. Κάθε φορά που εγώ έρχομαι σε επαφή ακόμα και με τους συναδέλφους από το Δημοκρατικό Κόμμα, το βρίσκω πολύ δύσκολο να το συζητήσουμε. Γιατί τελικά σε σχέση με τη δική μας συζήτηση, αυτοί βάζουν το κάρο πριν από το άλογο. <clears throat> δηλαδή ενώ εμείς λέμε εξυγίανση των οικονομικών και να δούμε τι θα γίνει μετά των δημοσιονομικών, αυτοί κάνουν το αντίθετο. για τους Αμερικανούς υπάρχει το πρόβλημα της μη βιώσιμης, της μη αηφόρου κατανάλωσης, του επίπεδου κατανάλωσης που οδηγεί σε προβλήματα στις παγκόσμιες ενισομέρειες. Μόνο με μια αλλαγή του μοντέλου διανομής μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η αλόγιστη υπερκατανάλωση από την πλευρά των Αμερικανών και από την πλευρά των Κινέζων έχουμε ένα διαφορετικό πρόβλημα αν θέλουμε να μιλήσουμε για σύστημα παγκόσμια διακυβέρνηση δεν θα συμμετάσχουν. Συμμετέχουν μόνο στο G20 γιατί δεν είναι δεσμευτική η απόφαση των G20. <clears throat> Επομένως το περιθώριο ελιγμών που έχουμε για να μπορούμε να παίξουμε κάποιο πολλαπλασιαστικό αποτελέσμα είναι πολύ περιορισμένο. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ. ανησυχώ δεν θα γίνει συζήτηση γιατί σε όλα συμφωνούμε, έτσι φαίνεται. Τέλος πάντων παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Το πρώτο θέμα είναι πώς ακριβώς θα συνενέσουμε, πώς θα επιτύχουμε ομοθυμία. Καταλαβαίνετε την απόγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συχνά γιατί προσπαθούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη για διάφορα ζητήματα και όχι μόνο στο πλαίσιο των συναντήσεων G20 αλλά και στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπαθούμε να τα πείσουμε να εισέλθουν σε ένα σύστημα ευρωπαϊκό ή άλλο όπου θα εκπροσωπούνται καλύτερα οι πολιτικές μας. Έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα προόδου αλλά ε, σίγουρα στο πλαίσιο της ομάδας G20 δεν είναι ιδανικά τα πράγματα, δεν είναι ιδανική η κατάσταση. Πολλοί Ευρωπαίοι ε, λειτουργούν και αντιπαραγωγικά συχνά. Τι γίνεται στην ομάδα G20, έχετε παραδείγματο χάρη τον ε, Βραζιλιάνο ή πώς να το πω τον Ιταλό που μιλάει μετά το Γερμανό και λένε όχι δεν σας ακούω πια γιατί όλοι τα ίδια λέτε Τέλος πάντων, ορισμένοι συμμετέχουν στο διάλογο με αντιπαραγωγικό τρόπο. και θέλω να καταλήξω. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση προσφέροντας έναν συντονισμό. Κάποιοι όροι terms of reference έχουν συζητηθεί με τα κράτη-μέλη γιατί δεν είναι Όλοι οι παρόντες στη συνεδρία της G20 εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εκπεριτροπής Προεδρία για ε, τους όρους αυτούς για τα Terms of Reference ε, συνεννοούμαστε εκ των προτέρων. Και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κάθε φορά τηρεί απαρέγκλητα αυτούς τους όρους επί των οποίων έχει συμφωνήσει με τα κράτη-μέλη και συντονίζουμε και τις ε, θέσεις της Ένωσης εκ των προτέρων. Δηλαδή, κάθε φορά που συνεδριάζει G20, ε, διαφορετικά επίπεδα κάθε φορά, προσπαθούμε να επιτύχουμε έναν συντονισμό των θέσεών μας εκ των προτέρων για να αποφύγουμε ακριβώς αυτές τις αντιδράσεις της Βραζιλίας ή οποιοδήποτε άλλο που λένε άμα όλοι τα ίδια λέτε και δεν γίνεται διάλογος. Προσπαθούμε να μιλούμε με μία φωνή ε, πάντως θα συμφωνήσω μαζί σας, ε, κυρία Περέσε, δεν ε, είναι ιδανική αυτή η μεθοδολογία. Πολύ καλύτερο θα ήταν να εκπροσωπείται από έναν μόνο, από ένα φορέα η Ένωση. Για την Ιαπωνία και πάλι θα συμφωνήσω μαζί σας. Το βασικό ελάττωμα, αν θέλετε, της λειτουργίας του G20 είναι ακριβώς η έλλειψη μηχανισμού υλοποίησης ε, των αποφασιστέντων. Εγώ είμαι Βέλγος. Γνωρίζετε πόσο καιρό, εδώ και πόσο καιρό παλεύει η χώρα να σχηματίσει η κυβέρνηση. Και την ίδια δυσκολία φαίνεται να αντιμετωπίζει και η Ένωση στις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα στα πλαίσια του G20. Πάντως, δεν συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι δεν μπορούμε να το στήσουμε ε, αυτό ε, το θέμα με τη ΣΥΠΑ, γιατί θα μας πούνε ε, από το Υπουργείο Οικονομικών, τον ίπα, ότι χτυπάτε την ανάκαμψη κατά αυτόν τον τρόπο, παρεμποδίζετε την ανάπτυξη και θα μας πούνε όχι θα πρέπει ποσοτικά να χαλαρώσετε λίγο τους όρους, να ακολουθείτε τις δικές μας μεθοδολογίες Τέλο πάντων, ναι, δεν υπάρχει σύμπνη απόλυτη. Έχουν την άποψή τους, έχουμε και εμεί τη δική μας ε, και προσπαθούμε να βρούμε μια φρασιολογία που συγκαλύπτει ε, ε, τη, τη διάσταση απόψεων, αλλά τουλάχιστον γίνεται διάλογος. Για την Κίνα και πάλι θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να να παίξουν το παιχνίδι όπως όλοι οι υπόλοιποι οι εκπρόσωποι της Κίνας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα στη Σεούλ, στην τελευταία συνεδρίαση. Ακόμη και με τους συναδέλφους με τους οποίους έχουμε σοβαρότατη διάσταση απόψεων, με προσώπους της Βραζιλίας, της Αργεντινής παραδείγματος χάρη, γιατί έχουν διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, προβάλλουμε εμεί την επιχειρηματολογία μα, εκείνη τη δική του και με το διάλογο προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα είδο συνένεση. Με του Κινέζου εκπροσώπου δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Εμεί παρουσιάζουμε τα επιχειρήματά μα και εκείνοι μα λένε όχι. Μην με ρωτήσετε πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Οι Αμερικανοί έχουν δοκιμάσει διάφορα συστήματα για τις σωτημίες. Ε, ε, προσπάθησαν με καλό τρόπο, με δημόσιο τρόπο, με ιδιωτικό τρόπο, με απειλές ε, στο Κογκρέσο, με διάφορους τρόπους προσπάθησαν να δώσουν μια απάντηση, αλλά τι, εγκρίθηκαν κάποιες νομοδοτήσεις και τίποτα άλλο, κάποια ψηφίσματα. Ε, προσπαθήσαμε από κοινού με τους Αμερικανούς ε, με ήπιο φιλικό τρόπο και λιγότερο φιλικό τρόπο να λύσουμε το ζήτημα. Δεν τελεσφόρησαμε το αυτές τις προσπάθειες. Φαίνονται κάπως πιο διαλλακτικοί ε, οι Κινέζοι, αλλά επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει τίποτα στην ισοτιμία εξαρτάται από την ημέρα, δηλαδή το ευρώ είναι λίγο, από, λίγο πάνω ή λίγο κάτω ε, σε σχέση με τα, την, ε, την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο. Ε, πάντως, όσοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα την Κίνα από μένα ενώ μου λένε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, χρειάζεται χρόνος. Είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, θα διακόψω για να πω το εξής οι Κινέζοι θέλουν να κάνουν την ε, Σανγκάη ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά, χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου. Για να το κάνουν αυτό πρέπει να γίνει το ρενμίμπι ένα βασικό νόμισμα μετατρέψουμε φυσικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό ή όχι. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που είμαι έτοιμος να συζητήσω στη δεύτερη φέτα συζητήσεων, στο δεύτερο τμήμα των συζητήσεων. Αλλά οι εμπειρογνώμονές μας στην Κίνα λένε ότι θα λειτουργήσει αυτό, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο καιρό, διότι οι Κινέζοι σκέφτονται σε αιώνες και χιλιετίες και όχι σε χρόνους και μήνες. Σας ευχαριστώ για την πλήρη σας απάντηση. Ο Γκίνορ Χέκμαρκ και μετά θα ακολουθήσει η Ελίζα Φερέιρα και σας παρακαλώ να απαντήσετε και στους δύο ομού και μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ βλέπω ότι όχι μονάχα χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό, αλλά χρειάζονται δύο και για μια ανισομέρεια. Το ξεχνάμε αυτό, γιατί όταν μιλάμε για ανισομέρειες, μιλάμε για τους άλλους. Για τα προβλήματα που δημιουργούν οι άλλοι, για τις ανισομέρειες των άλλων. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πάντα, έτσι το βλέπουμε. Αλλά αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για ισοτιμίες σε άλλες ε, περιπτώσεις. Έχω κάποιες επιφυλάξεις λοιπόν για μια προσέγγιση η οποία αφορά περισσότερο τους άλλους και όχι εμάς τους ίδιους. Αυτό είναι λίγο παράξενο ακόμα και για ταγκό. Μερικές φορές μου λείπει να υπάρχει μια περισσότερη προβληματική για το γιατί υπάρχουν αυτές οι παγκόσμιες ανισομέρειες. <clears throat> και πρέπει να σκεφτούμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ότι και εμείς αφήσαμε πίσω μας ορισμένες ανισομέρειες. Αν πάρουμε τα τελευταία 20-25 χρόνια που περάσανε. Η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει εκ βάθρων. Έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε σχετική ευμάρεια από 1 σε 4 δισεκατομμύρια. Και έχει μειωθεί η ένδια σε ένα αδιανόητο σχεδόν επίπεδο σήμερα. Βέβαια, οι τεράστιε ε, ανισότητες που υπήρχαν τότε δεν τις καταλαβαίναμε γιατί είχαμε τον κόσμο χωρισμένο σε τρία οικονομικά στρατόπεδα. Πρώτος κόσμος, δεύτερος κόσμος, τρίτος κόσμος. Και το τι γινόταν εκεί κάτω δεν μας απασχολούσε. Τώρα έχουμε μια νέα παγκόσμια οικονομία με νέες παγκόσμιες ισορροπίε ή ανισορροπίε, καλύτερα για να το πω έτσι. Και ένα από τα κυριότερα προβλήματα σε αυτή την παγκόσμια ισορροπία και ανισορροπία είναι ότι <clears throat> εμείς δεν έχουμε προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Βλέπουμε να υπάρχουν αυτά τα ελλείμματα στις, στα δημόσια οικονομικά και στο να υπάρχει και σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη έχουμε τέτοια ελλείμματα γιατί καταναλώνουμε περισσότερο από ό,τι παράγουμε. Μακροχρόνια είναι ένα πρόβλημα δεν μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση για τις παγκόσμιες ισορροπίες και μη ισορροπίες να τεθεί σε μια ευρύτερη ισορροπία και όχι μονάχα με γνώμονα το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και τα δημοσιονομικά. Δεν υπήρξε καμιά συζήτηση για το εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο, γιατί αυτά τα οποία είδαμε στις δύο-τρεις τελευταίες δεκαετίες είναι η τεράστια ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου με θετικές επιπτώσεις που προέκυψαν. Αλλά ήταν ασυμμετρική ανάπτυξη σε όλα αυτά. Γιατί η Γεωργία δεν έχει υπαχθεί στην πλήρη παγκοσμιοποίηση, ούτε οι περισσότερες υπηρεσίες. Και οι περισσότερες υπηρεσίες είναι προς όφελος της ευρωπαϊκής και αμερικανικής οικονομίας και τα περισσότερα προβλήματα, αν υπάρξει πλήρης απελευθέρωση του παγκοσμίου εμπορίου, θα, αυτή η απελευθέρωση φιλελευθεροποίηση θα είναι προς όφελος του τρίτου κόσμου, όπου υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για εξαγωγές. Αναρωτιέμαι λοιπόν, Έχετε κοιτάξει το θέμα του ελεύθερου εμπορίου και τις επιπτώσεις στις ε, ανισομέρειες αυτές. Γιατί αυτό θα επηρεάσει τα πάντα, σε, όλες τις, ε, σε όλα τα επίπεδα της ανισομέρειας. Η κυρία Φερέα, μπορώ να μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα έθετα το εξής ερώτημα, λοιπόν. Όταν ε, μιλάμε για την κρίση, ε, ε, θεωρούμε ως δεδομένο ότι όλος ο κόσμος ζει μια κρίση. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Χόκμαρκ μόλις τώρα, έχουμε μια κρίση στην Ευρώπη και μια άλλη στη ΣΥΠΑ. Ε, στον ε, υπόλοιπο κόσμο ε, υπάρχει μια μικρή φεσούλα σε σχέση με την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών. Οπότε τώρα τι, ποιο θέμα εξετάζουμε, ποιο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το νέο κόσμο, σε αυτή τη νέα εποχή στην οποία έχουμε περάσει. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι έχουμε μια συνταγή για τη ΣΥΠΑ, μια συνταγή για την Κίνα, αλλά η συνταγή για την Ένωση είναι συγκεχημένη, ε, διότι αν δείτε τις ανισορροπίες ε, στις τρέχουσες ε, συναλλαγές, βλέπουμε στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο χώρος όπου δεν υπάρχει μεγάλη ανισότητα είναι ακριβώς η ζώνη ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο ως προς τις εμπορικές συναλλαγές η ΕΠΑ και η Κίνα είναι δύο εμπορικοί εταίροι αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια σχετική ισορροπία. Δηλαδή μπορεί να ε, αναλάβει αν θέλετε και ηγετική θέση η Ένωση άμα πιστέψει κάποιο το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα δεν είναι αλήθεια αυτό γιατί υπάρχει θεσμικό ζήτημα. Αν δεν έχουμε σε θεσμικό έρισμα δεν γίνεται να αναλάβει τέτοιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυρίω επειδή βρίσκεται σε επισφαλή θέση λόγω άλλου είδου ε, ανισοτήτων και αυτές πρέπει να τις συζητήσουμε. Ε, και θεωρώ ότι τρεις, τρεις διάστατες είναι αυτές οι ανισότητες. Πρώτον, ε, ανεπαρκής οικονομική ανάπτυξη. 1% ανάπτυξη φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας, δεν επαρκεί. Οπότε η αναπτυξιακή πολιτική είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Ίσως όχι τώρα εδώ, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στη στρατηγική 2020 γιατί δεν έχει επαρκή κονδύλια ούτε και τα απαιτούμενα μέσα. Δεν έχουμε ανεπτυξιακή πολιτική ουσιαστικά. Δεύτερον, ε, το δημόσιο χρέος ε, ε, και που όλες οι άλλες δυσκολίες που προκύπτουν από το ενιαίο νόμισμα και δημιουργούν προβλήματα στις χώρες που συναποτελούν τη ζώνη ευρώ. Οπότε η συνταγή διόρθωσης της ε, ανισορροπίας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι αυτή που προτείνει η ομάδα G20, δεν μπορεί να είναι η απάντηση μόνο η δημοσιονομική εξυγίανση που πλήττει ε, την ανάπτυξη. Το αντίθετο, οι χώρες που κάνουν τη δημοσιονομική οικονομική εξυγίανση κοντόθαλμα εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Μέσω μακροπρόσμα δεν έχουν καμία πολιτική που θα εξασφαλίσει την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Αυτά τα συστήματα, αυτά τα θέματα είναι αρκετά σημαντικά ώστε να συζητηθούν τώρα. Αλλιώς θα απολέσουμε τον έλεγχο, θα απολέσουμε το ρόλο που μπορεί σε διεθνή κλίμακα να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, ε, κάθε ένας από αυτούς τους φορείς έχει τη δική του εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν έχει σαφή ε, εξωτερική εμπορική πολιτική. Για το fair trade ε, ε, πρέπει να παλέψουμε για το ίσο εμπόριο, όχι για το free trade, το ελεύθερο εμπόριο. Δεν μπορούμε να δίνουμε ασαφή μηνύματα δηλαδή αυτός ο εξωτερικός εμπορικός ε, φραγμός ε, που υπάρχει είναι ασύμετρος ε, και πλήττει με διαφορετικό τρόπο τις χώρες, επιμέρους χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank you. Um, I'll try to, to speak. Θα προσπαθήσω να διεξέλθω τα ερωτήματά σας με τη σειρά που τα διατυπώσατε. Κάποια από τα ερωτήματά σας νομίζω ότι ήταν παρόμοια, γιατί αναφερθήκατε και οι δύο στο γεγονός ότι μιλάμε για το τι θέλουν να κάνουν, θέλουμε να κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν λέμε τίποτα για αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Δεν συμφωνώ βέβαια απόλυτα, γιατί εγώ παρουσίασα ορισμένα στοιχεία της σκέψης μας, αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η δική μας συμβολή στη μείωση των παγκοσμίων ανισομεριών Μίλησα για την Ευρώπη 2020 που δεν είναι βέβαια επαρκής από μόνη της αυτή η στρατηγική. Ο κύριος τώρα λόγος για τον οποίο δεν, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες για το τι πρέπει να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τις παγκόσμιες ανισομέρειες είναι, όπως είπε η κυρία Φιρέιρα, ότι εμείς δεν συμβάλλουμε τόσο πολύ στις παγκόσμιες ανισομέρειες το, η θέση της Ευρωπαϊκής ε, ε, της ζώνης του ευρώ σε επίπεδο ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι περίπου ισοσκελισμένη, ισορροπημένη και προβλέπεται να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούμε να πράξουμε πολλά για να μειώσουμε τις παγκόσμιες ανισομέρειες, ακριβώς γιατί η πηγή αυτών των ανισομεριών δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη ζώνη του ευρώ. Αδειρήτως λοιπόν η εστίασή μας θα πρέπει να τεθεί στους άλλους το πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτοί. Μήπως λοιπόν το άλλο ερώτημα πως θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη αντιμετώπιση και όχι να περιοριστούμε στο ισοζύγιο τρέχουσων πληρωμών. Βέβαια μπορούμε να το κάνουμε. Όταν μιλάμε μεταξύ οικονομολόγων και λιπτών αποφάσεων στους G20, αυτά λέμε. Λέμε και άλλα πράγματα πέραν του ισοζυγίου τρέχουσων πληρωμών. Αλλά οι Κινέζοι, γιατί για τους Κινέζους πρόκειται, όταν δακτυλοδεικτούσαμε την Κίνα και λέγαμε εσείς συμβάλλετε στην ανισομέρεια ε, του ισοζυγίου πληρωμών λόγω του υποτιμημένου σας ρεμβιμβίου λέγανε οι Κινέζοι και άλλε ανισομέρειε η διαφορά μεταξύ των φτωχών περιοχών στην Κίνα και των πλουσίων, οι ανισομέρειε μεταξύ Αφρική και, προχωρη... και προκεχωρημένων οικονομιών και αυτό δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Για αυτού ήταν ένα τρόπο να αγνοήσουν το πρόβλημα και να μην συμβάλλουν στη γενική συζήτηση. Από έποψη τακτικής λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ίσως καλύτερο να δώσουμε προσοχή και έμφαση στην, ε, στα θέματα ισοζυγίου πληρωμών, ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών, συγγνώμη, και όχι να καλύψουμε όλο το φάσμα των προβλημάτων. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε τίποτα με τους Κινέζους. Θέλετε να επανέλθετε. Ναι, ναι, για περισσότερη σαφήνεια. Αυτό το οποίο έλεγα εγώ δεν είναι ότι θα πρέπει να συζητήσουμε άλλες ανισομέρειες, αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά προβλήματα θα πρέπει να δούμε και τις μακροχρόνιες εξελίξεις οι οποίες προεκλήθησαν από αυτούς τους παράγοντες. Και θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε στις νέες πραγματικότητες. Αυτό ήταν περισσότερο το τι ήθελα να πω. Συμφωνώ. Υπάρχουν πολλά θέματα που είναι η ρίζα του προβλήματος που καταδίονται πολύ πιο σε βάθος σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε. Αναφερθήκατε και στο εμπόδιο, στο εμπόριο, όχι στο εμπόδιο, συγγνώμη. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα. Είναι κάτι το οποίο επανέρχεται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση των G20 ότι πρέπει να κάνουμε πρόοδο σε σχέση με, τις, με την εφαρμογή των ε, συμπερασμάτων του γύρου της ΔΟΧΑ. Και ως Ευρωπαίοι εμείς θέλουμε να προωθήσουμε αυτά τα συμπεράσματα αλλά η εντύπωσή μας είναι ότι κάποια άλλα τμήματα του κόσμου οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται εξίσου στην εφαρμογή αυτών των συμπεράσματων και για τη γεωργία. Θέλω το δικηγόρο μου για να μπορέσω να μιλήσω, αλλιώς δεν λέω τίποτα. Για αυτά που είπε η κυρία Φιρέιρα, θα συμφωνήσω ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε τις ε, ανεπτυγμένες οικονομίες και χώρες ε, όπως αυτές που βλέπουμε συνέχεια στον τύπο, την Ισία, Αίγυπτος ε, δεν επλήγησαν γιατί ήταν ε, σχετικά προφυλαγμένες από τις εξωτερικές εμπορικές ε, ε, συναλλαγές, ήταν κλειστές οικονομίες δηλαδή. Αυτές οι πολιτικές βέβαια δεν μπορούν να συνεχίσουν να ακολουθούν αυτή την πολιτική με αυτή αυτό το πρόσχημα ότι εφόσον δεν πληγήκαμε από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο για να προστατευτούμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει τα είπαμε και προηγουμένως αυτά, αλλά εσείς αναφερθήκατε συγκεκριμένα σε τρία επιμέρους σημεία για το μελλοντικό ρόλο της Ένωσης. Go Όπως σας είπα και στην αρχή, έχω πολύ πιο καλά κατρετισμένους συνάδελφους και θα μπορούσα να σας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις όταν γίνουν ε, συζητήσεις ειδικά για αυτά τα θέματα, για εγχώρια ζητήματα αν θέλετε. Εντάξει, αυτά που είπατε για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι θα λύσει όλα τα διαρθρωτικά μας προβλήματα. Μάλλον υπερβάλλουν όσοι το ισχυρίζονται κατά ε, λίγο. Αλλά τι να σας πω άλλο. Νομίζω ότι απάντησα στην κυρία Φερέιρα. Ο κύριος Όλε Σμίτ και μετά ο κύριος Σβόποντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν όπως λέτε το πρόβλημα είναι ότι οι προαναφερθήσεις χώρες επαναλαμβάνουν ε, και μένουν στη θέση τους, ε, δεν βλέπω το πρόβλημα, αλλά ε, για να το πω πιο συγκεκριμένα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική στάση. Δηλαδή αυτές οι τέσσερις-πέντε χώρες να εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λύσουμε έτσι το πρόβλημα. Εσείς ε, σήμερα εκπροσωπείτε τη γυραιά Ήπειρο. Ε, στο μέλλον μπορεί ε, να μην ισχύει αυτό. Ίσως θα έπρεπε ε, να φανούμε λίγο ευφιέστεροι για να λύσουμε όλα αυτά τα σοβαρότατα προβλήματα. Η ομάδα G20 παρότι ε, υπάρχουν οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου μέσα στη G20 παρόλα αυτά πολλοί δεν εκπροσωπούνται σε αυτήν την ομάδα. Αυτό το συζητάτε καθόλου πώς θα πώς θα εκπροσωπηθούν αυτές οι χώρες, πώς θα, έχουμε μία, πώς, πώς θα μιλάμε όλοι με μια φωνή και θα φτιάξουμε ένα παγκόσμιο σύστημα εάν δεν εκπροσωπούνται στην G20 τόσες πολλές χώρες. Δεν πρέπει να δώσετε και μια απάντηση σε αυτό. Τώρα για την Κίνα. Κάνατε κάποια σχόλια σε σχέση με τι πρέπει να κάνει η Κίνα, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πρέπει να κάνει η ομάδα G20. Αλλά γιατί δεν μιλάτε για το πολυκομματικό σύστημα και για τη δημοκρατία καθόλου. Ε, είναι αδύνατον ε, να εκδημοκρατιστεί η Κίνα ε, στους Financial Times πριν από λίγες εβδομάδες πολλά δημοσιεύματα έλεγαν ουσιαστικά ότι η έλλειψη δημοκρατία στην Κίνα είναι εποφελής για την χώρα η έλλειψη των δημοκρατικών θεσμών. Αν κάνετε μία αντιπαραβολή με την Ινδία θα διαπιστώσετε ότι εκεί πολύ δυσκολότερα θα λύνονταν αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα. Τέτοιου είδους ζητήματα συζητιούνται στο G20. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Τώρα τέλος ε, ε, για τη Σαουδική Αραβία. Όταν μιλάει η Σουηδική Αραβία, τι ε, εκπροσωπεί τον Αραβικό Σύνδεσμο, τις αραβικές χώρες, τις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο και πώς το συνδυάζεται αυτό με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική η στάση της Σαουδικής Αραβίας ε, και στα πλαίσια του G20 στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η τωρινή κατάσταση βέβαια είναι συνδυασμός δομικών ανισομεριών που είχαμε εδώ και πολύ καιρό και της χρηματοπιστωτικής κρίσης η οποία ήλθε και προσθέθηκε σε αυτά. Υπάρχει αυτή η έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου για την κρίση που βγήκε πριν από ορισμένε μέρες την έχει μελετήσει η Κομισιόν, έχει πάρει κάποια θέση η Κομισιόν για τα συμπεράσματα αυτή της έκθεσης. Δεν φαντάζομαι τώρα ότι θα υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς τη βλέπει η Κομισιόν αυτή την έκθεση. Δεύτερον, για τους G20 να επανέλθω σε αυτό το οποίο ελέγχθη και μπορούμε να το συνδέσουμε και με το επόμενο σημείο αποτελεσματικότητα. Εντάξει, η δημοκρατική λογοδοσία είναι κάτι σημαντικό για αυτόν τον ιονή οργανισμό. Δεύτερο όμως είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, πόσο αποτελεσματική είναι. Κωστής της Παναγιάς στα μάτια, προκαλεί διαδηλώσεις, πέφτει ξύλο, τα μέσα ενημέρωσης ε, ασχολούνται, αλλά στην πράξη τι προκύπτει από όλα αυτά. Μήπως σκέφτεται η Κομισιόν να υπάρξει κάποιος τρόπος να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η συνεδρίαση ή να ενσωματωθούν οι G20 σε κάποιο ευρύτερο φορέα. Ποια είναι η θέση g Κομισιόν. Και επίσης η αλληλοσύνδεση μεταξύ των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών προβλημάτων. Το θέμα της κερδοσκοπίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο θέσεις. Τουλάχιστον φραστικά αυτά τα οποία είπε ο Σαρκοζή που είπε ότι η κερδοσκοπία έχει παίξει ένα τεράστιο ρόλο, ενώ η Κομισιό λέει όχι, η κερδοσκοπία δεν έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Εσείς στην έκθεσή σας για τη βιομηχανία και τα βασικά προϊόντα παρουσιάσατε την κατάσταση που είναι διαφορετική βέβαια. Πού θα καταλήξουμε, θα πείσετε τον Σαρκοζή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κερδοσκοπία στα βασικά προϊόντα, ο Σαρκοζή θα σα πείσει ότι δεν υπάρχει κερδοσκοπία ή θα βρεθείτε στο δρόμο τη Καμίλα, στη μέση δηλαδή. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η θα βρεθειτε στον δρομο δεν είναι αυτή η οποία οδηγεί σε ανισομέρειες. Ίσως η κερδοσκοπία να συμβάλλει σε κάποιο βαθμό στην ενίσχυση κάποιων ανισομεριών. Και όλα αυτά με ξαναφέρνουν στο πρώτο ερώτημα το οποίο ετέθη. Αν η κερδοσκοπία ενισχύει και οξύνει τις ανισομέρειες, το ερώτημα είναι αν έχουμε καλύψει όλο το δρόμο της επαναφοράς της ρύθμισης ή όπως λένε οι Αμερικανοί πρέπει να δημιουργηθεί ένα επιπλέον παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο όχι με την ε, παλιά έννοια της δεκαετίας του 40 αλλά με τη νέα σύγχρονη αντιμετώπιση. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Για το αν μιλάμε με μία φωνή ή αν επαναλαμβάνει ο ένας και επικαλύπτει τον προηγούμενο. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να έχουμε ένα απλούστερο σύστημα στα πλαίσια των οποίων να εκφράζονται τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν τα μεγάλα κράτη-μέλη το θέλουν αυτό. Γιατί αν η Γερμανία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν εκπροσωπεί ουσιαστικά τη Γερμανία, λέει ο μιλητής. Και στην ουσία μειώνεται κατά πολύ ο αριθμός και το πεδίο, αν θέλετε, της αναφοράς για κάθε μία χώρα. Όταν εμείς συζητάμε όμως το θέμα σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν αναλύουμε τις πιθανές συνέπειες της συνθήκης της Λισαβόνας σαν παράδειγμα, βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ομάδας των 20, όχι σε επίπεδο ηγετών, γιατί εκεί Υπάρχει ήδη συμφωνία για τον Παρόσο ή τον Βον Ρόμπαϊ. Αλλά σε επίπεδο θα έλεγα χαμηλότερο θα μπορούσε να είναι είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε ένας ειδικό απεσταλμένος είτε η κυκλική προεδρία. Το θέμα όμως παραμένει αυτό που είπα στην αρχή. Οι μεγάλες χώρες μέλη το θέλουν αυτό υπάρχει μια γενικότερη θεωρητική συζήτηση γύρω από την αντιπροσωπευτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ομάδας των 20. Εδώ υπάρχει ένα αντιστάθμισμα ανάμεσα στα δύο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Θελήσατε να μάθετε αν συζητιέται και συζητιέται. Θεωρείται η ομάδα των 20 ότι δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Η ίδια λοιπόν εσωτερικά θέλει να είναι αντιπροσωπευτική. Η Κορεατική Προεδρία, σαν παράδειγμα, έδωσε την δυνατότητα στο Μαλάουι να πάρει μέρος σε πολλές συναντήσεις, στην Αιθιοπία, στη Σιγκαπούρη. Περιοδικά γίνονται αυτά τα ανοίγματα έτσι ώστε να φανούμε δεκτικοί σε χώρες εκτός της ομάδας των 20. Είναι κοινό τόπος δηλαδή ότι οι χώρες αυτές οι οποίες βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή θα πρέπει να επικοινωνούν με τις όμορες χώρες για το τι συμβαίνει στην ομάδα των 20. Η Νότια Αφρική θεωρεί ότι έχει συγκεκριμένο ρόλο ενημερώνοντας, πληροφορώντας την λεγόμενη υποσαχαρική Αφρική για τα τεκτενόμενα στην ομάδα των 20. Σαουδική Αραβία το ίδιο κάνει και για τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου. Τώρα για το αν αντιπροσωπεύουν τον Αραβικό Σύνδεσμο οι Σαουδάραβες ή τις πετρελοπαραγωγές χώρες. Η Σαουδική Αραβία όταν εκφράζεται περισσότερο εκφράζεται μέσω θα έλεγα των πετρελοπαραγωγών χωρών. Περισσότερο και ίσως αμέσως μετά να έρχεται η αντιπροσώπευση από πλευρά της της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι γενικότερα, ειδικότερα του Αραβικού Συνδέσμου. Τώρα, για την αποτελεσματικότητα και το υπόλογο σε εισαγωγικά της ομάδας των 20. Η ομάδα των 20 είναι ήδη μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πολλές φορές έχει κανείς την αίσθηση ότι οι συζητήσεις κρατάνε πάρα πολύ οι συζητήσεις δεν είναι ουσιαστικές συζητήσεις, είναι διαδοχή δηλώσεων, δεν γίνεται αρκετή, δεν υπάρχει διαδραστικότητα και πολλοί θέλουν να μειώσουν το μέγεθος αυτής της ομάδας για να υπάρχει μεγαλύτερη διαδραστικότητα, αλληλοεπίδραση και καλύτερα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εγώ δεν δίνω λύσεις. Οι λύσεις που δίδονται είναι η δημιουργία ομάδων μικρότερων, ομάδων εργασίας, υπο-ομάδων τομέων. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί κανείς να σπάσει τις συζητήσεις ε, επιμέρους θεματικά, αλλά και αυτό απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Πρακτικά λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας, συγγνώμη. Και εδώ έρχομαι με αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Βόμποντα, το οποίο ρώτησε ο κύριος Βόμποντα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων της ομάδας των 20. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη ομάδα. Υπάρχει πάντα, θυμίζω, η ομάδα των 8. Υπάρχει πάντα η ομάδα των 7. Κάτι λέει η κυρία Μπερές εκτός μητροφώνου δεν ακούμε. Στο Τορόντο είχαμε συνεχείς εφαπτώμενες συναντήσεις της ομάδας των 8 και της ομάδας των 20 και υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι πήραν μέρος και στις δύο συναντήσεις και είπαν ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το G8 έχει διαλυθεί πλέον, τερμάτισε και ότι το G20 το διαδέχθη. Λοιπόν, έτσι πιστεύουν ορισμένοι. Δεν υπάρχει όμως, επαναλαμβάνω, εφαρμοστικός μηχανισμός των αποφάσεων της ομάδας των 20. Εν πάση περιπτώσει. Η επιρροή του ενός στον άλλο παίζει κάποιο ρόλο. Και όταν υπάρχει μια κάποια συμφωνία, τουλάχιστον αν δεν εφαρμόζουν τη συμφωνία, προσπαθούν να την, να την εφαρμόσουν. Υπάρχει δηλαδή μια κίνηση προς τα εκεί. Και θυμίζω ότι η ομάδα των 20 ήταν σχετικά αποτελεσματική καταπολεμώντας την οικονομική κρίση. Όταν ξέσπασε η κρίση υπήρξε ένα συντονισμό των προσπαθειών σε πλαίσιο G20 και οι χώρες εφήρμοσαν αυτά τα οποία τους ζήτησε το G20. Τώρα υπάρχει αίσθηση ότι βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση. Δεν ήταν εύκολη η κρίση αυτή, ήταν τεράστια, αλλά ταυτόχρονα όλοι είχαμε τα ίδια συμφέροντα και τους ίδιους στόχους. Ως εκ τούτου ήταν εύκολο να εφαρμόσουμε τα αποφασισμένα. Τώρα όμως διαφοροποιούνται οι στόχοι. Οπότε είναι πιο δύσκολο κάποιες χώρες να εφαρμόσουν αυτά τα οποία αποφασίζονται σε επίπεδο G20. Υπάρχει όμως όπως είπα ε, μια προσπάθεια αντιστάθμισης ισορροπίας. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς αν οι αποφάσεις λαμβάνονται, που λαμβάνονται σε επίπεδο G20 είναι πιο αποτελεσματικές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε G8. Ίσως θα πρέπει να τα σπάσουμε σε μικρές ομάδες. Κάποιοι ας πούμε οι Κινέζοι επιμένουν ότι το βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητάμε είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, κάποιοι άλλοι όχι. Τώρα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανεξάρτητη άποψη, όχι δεν τίθεται έτσι το θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται συνεχώς. Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα πρόταση, ξέρουμε ας πούμε ότι η κυρία Λαγκάρντ είναι ιδιαίτερα παραγωγική, κάνει προτάσεις εμείς αναλύουμε τις προτάσεις αυτές, εκφέρουμε άποψη πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το πώς βλέπουμε αυτές τις προτάσεις. Αυτό το οποίο πρέπει όμως είναι η Ευρώπη να καταφέρνει να εκφράζεται με μία φωνή. Έτσι ώστε οι ασδήποτε αλλαγές ε, ε, διαπιστώνεται ότι είναι χρήσιμο να γίνουν οι αλλαγές αυτές να μπορούν να εφαρμοστούν με ενιαίο τρόπο και γι' αυτό οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβώς αυτές που ε, ε, είναι προτάσεις που συνδυάζουν τις προτάσεις που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Βέβαια η προσπάθεια είναι τεράστια. Ε, δεν έχουμε όλους τους πόρους σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνουμε τις αναλύσεις οι οποίες απαιτούνται αλλά δεν είναι κάτι εύκολο για μας. Προσπαθούμε. Ευχαριστώ. Εμείς είχαμε συναντήσει στις ΗΠΑ τον πρόεδρο της ομόλογου επιτροπή μας με τους συνεργάτες τους και είχαμε συμφωνήσει ότι όταν τελειώσει με την έκθεσή του θα μας την ε, δώσει και εμάς. Είμαστε λοιπόν σε επαφή για να δούμε αν αν θα υπάρξει κοινή στάση στην έκθεση αυτή. Έχουμε έξι δημοκράτες οι οποίοι έχουν υποστηρίξει αυτή τη στιγμή την έκθεση, ενώ οι τέσσερις ρεπουμπλικάνοι είναι τρία προς ένα κάπως, δεν είναι ενωμένοι ούτε αυτοί, έχουν διαφορές απόψεων. Θα δούμε στη συνέχεια ποια θα είναι η άποψη που θα δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, ναι συγγνώμη. Ναι, ναι, υπήρχε κάτι το οποίο... Εγώ είπα κερδοσκοπία, εσείς είπατε Σαρκοζή. Υπήρχε αυτό το σημείο το οποίο έπρεπε να απαντήσω. Το αν η κερδοσκοπία παίζει κάποιο ρόλο ή όχι στην αγορά βασικών προϊόντων ιδιαίτερα ή αν δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα. Για το ελληνικό κρατικό χρέος κάτι ρωτήσατε. Ναι, ίσως αυτό έχει παίξει κάποιο ρόλο εδώ η κερδοσκοπία για το ελληνικό κρατικό χρέος. Η θέση της Κομισιόν ότι η κερδοσκοπία δεν αποτελεί πρόβλημα καθόλου. Εμείς έχουμε μια πιο επιφυλακτική στάση γιατί αυτό το οποίο λέμε είναι ότι μέχρι στιγμής φάση των αναλύσεων που έχουμε κάνει και δεν είναι τελείως περατωμένες και χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να καταδείξουμε ότι η κερδοσκοπία έχει παίξει κάποιο ρόλο. Αυτό είναι διαφορετικό από το να πούμε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο η κερδοσκοπία. Μπορούμε ακόμα να φτάσουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Επίσης θέλω να σα πω ότι η κερδοσκοπία μπορεί και σίγουρα να οξύνει τις χρηματοοικονομικές κρίσεις, αλλά μπορεί και να τις καταπραίνει και να μειώσει την έντασή τους. Εάν η κερδοσκοπία ουσιαστικά εξυπηρετεί την αντιστάθμιση κινδύνων εναντίον των μεγάλων διακοιμάσεων, αυτό έχει ένα καταπραγητικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε λοιπόν όλα τα κακά του κόσμου να τα αποδίδουμε στους κακούς κερδοσκόπους. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι δεν έχουμε ακόμα σταθμίσει απόλυτα τη θέση μας. Γίνεται η επεξεργασία και η ανάλυση και προς το παρόν δεν έχουμε ε, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει παίξει ρόλο η κερδοσκοπία. Φυσικά όλα αυτά θα συζητηθούν περισσότερο. Ο Νικόλαος Χούντης και η Ντανούτα Χούπτερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπέξ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρχική εισήγηση που κάνατε και επειδή μου δώσατε την εντύπωση πως έχετε αίσθηση του χιούμορ θέλω να σας πω ότι σας παρεξήγησα διότι στην αρχική εισήγηση διέκρινα αρκετή αισιοδοξία σε σημείο ενδεχομένως και αφέλειας. Βέβαια μετά στις απαντήσεις σας μοιάζεται να το βλέπετε πιο ρεαλιστικά τα πράγματα αλλά επιτρέψτε μου να ξαναπώ δυστυχώς το τελευταία απάντηση για την κερδοσκοπία και για το ελληνικό χρέος πάλι μου το χαλάσατε το θέμα. Εν πάση περιπτώσει σας εύχομαι να είστε αισιόδοξο, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Από πού υπάρχει, μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η προσπάθεια ενός μηχανισμού πρόβλεψης ή εξισορρόπησης αυτών των ανισορροπιών μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Ή να σας το πω πιο απλά, γιατί μια τα βάζουμε με την Κίνα, μια πλεονασματική χώρα θα δεχτεί κάποια στιγμή να μειώσει τα πλεονάσματά της. Εδώ έχουμε στην Ευρώπη, εδώ έχουμε στην Ευρωζώνη την πλεονασματική Γερμανία, η οποία δεν δέχεται να κάνει μια τέτοια κίνηση σε ένα πλαίσιο πιο δεσμευτικό από το πλαίσιο των G20 εν πάση περιπτώσει της παγκόσμιας συζήτησης. Και δεν πρόκειται να την κάνει αυτή την, την κίνηση. Ήδη βλέπουμε να την κάνει αυτή την κίνηση. Από πού λοιπόν προκύπτει αυτή η αισιοδοξία ότι οι πλεονασματικές χώρες κάποια στιγμή, και μιλώ ε, για την περίπτωση της Γερμανίας, γιατί και στη διεθνή συζήτηση, αν την έχω παρακολουθήσει καλά, υπάρχει ένας ανταγωνισμός Κίνας-Γερμανίας, ποια θα ξεπεράσει την άλλη η πρώτη έχει ξεπεράσει τη Γερμανία σε εξαγωγές αν δεν είμαι καλά ενημερωμένος. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τη δική μου διάθεση. Γιατί εγώ εξακολουθώ να είμαι απεσιόδοξος κύριε Μπέξ. Σε ποιο κομμάτι. Διότι αυτές οι ανισοτιμίες οφείλονται σε ανισορροπίες στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας των χωρών ή και των διαφόρων ε, ενωτήτων. Εκεί από αυτή την υπόθεση της ανταγωνιστικότητας διακρίνω συνεχώς στην ευρωπαϊκή πολιτική να δουλεύουμε μόνο με τη μεταβλητή που λέγεται κόστος εργασίας. Δηλαδή, οι πολιτικές που ακολουθούνται, αυτό που είπατε και η οικονομική διακυβέρνηση, κατά την άποψή μου, είναι μια συνεχής προσπάθεια κινεζοποίησης, να το πούμε έτσι, της κατάστασης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελαστικοποίηση των σχέσεων, ε, εργασιακών σχέσεων, μείωση των μισθών, ακύρωση του ρόλου των συνδικάτων, προκειμένου να κερδίσουμε σε ανταγωνιστικότητα. Πείτε μου σας παρακαλώ, να συνεχίσω να είμαι απεσιόδοξος ότι όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η συζήτηση, όταν δεν είναι αφελής, έχει αυτό το στόχο, δηλαδή μια ανταγωνιστικότητα που να προκύπτει μέσα από τη μείωση των δικαιωμάτων των μισθών, μέσα από σκληρά δημοσιονομικά προγράμματα λιτότητας, ενώ τα άλλα μένουν σε επίπεδο ευχολογίου και μια συζήτηση θα μπορούσε να πει κανεί ευχάριστη στα αυτιά αλλά όχι πραγματική όσο αφορά την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην ευρωπαϊκή ένωση. Thank uh, ε, Κυρία Χούμπνερ, συγγνώμη, δεν μπορούσα να με παρούσα για την παρουσίασή σας. Αλλά όταν μπήκα λέγατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στο ισοζύγιο τρεξών πληρωμών στην περίπτωση της Κίνας. Αυτό μου φαίνεται με ένα σωστό, εφόσον βέβαια δεν κοιτάμε την προσαρμογή ισοτιμιών ως το μόνο μηχανισμό για να αντιμετωπίσουμε τις ανισομέρειες. Νομίζω θα ήταν πραγματικά σφάλμα από την ευρωπαϊκή πλευρά εάν δεν βλέπαμε το σύνολο των διαρθωτικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που θα δημιουργήσουν ανισομέρειες στο μέλλον αλλά ελπίζουμε ότι ότι οι ανισομέρειες θα υπάρχουν στο μέλλον θα βασίζονται σε διαφορετικές ανταγωνιστικότητες και όχι σε υποτιμημένα νομίσματα. Είναι λοιπόν πάρα, πολύ ενδιαφέρον να δούμε το θέμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε συνάρτηση με τις εμπορικές ροές και με την, ε, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Μπορούμε όμως να το κοιτάξουμε και πιο πολύ σε βάθος γιατί αλλιώς μπορούμε να καταλήξουμε σε λανθασμένα ε, συμπεράσματα αν δεν κατανοήσουμε τις δομικές αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα και εξάλλου θα είναι πολύ πιο δύσκολο για μας να βρούμε ένα μηχανισμό προσαρμογής εάν οι Κινέζοι μπορέσουν να αποκτήσουν ένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όχι μόνο επί τη βάση των ισοτιμιών. Το ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω είναι το εξής βλέποντας την ανάλυση της Κομισιόν και αυτά που είπατε και εσείς και τις άλλες δυνάμεις οι οποίες παίζουν κάποιο ρόλο στα θέματα αυτά, βλέπουμε κάποιο αντίκτυπο που μπορεί να προκαλέσει από τις δυνάμεις αυτές κάποιες περαιτέρω ανισομέρειες στην παγκόσμια οικονομία στο μέλλον. Um, Οφείλω να διευκρινίσω κάτι. Όταν μίλησα για την κερδοσκοπία και είπα ότι δεν έχουμε καμία ένδειξη σχετικά με το ρόλο της κερδοσκοπίας. Αναφερόμουν στις εξελίξεις, στις τιμές ε, των τροφίμων και των βασικών εμπορευμάτων και όχι στην Ελλάδα. Ε, δεν αναλύσαμε το πώς επηρεάζει η κερδοσκοπία τι ελληνικές ε, χρηματοπιστωτικέ αγορές και αν λόγω της κερδοσκοπία συμπεριφέρθηκαν με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Ε, σχετικά με το αν ε, είμαστε αφελείς, αισιόδοξοι και προσπαθούμε να μεταπίσουμε τους Κινέζους, θα σας απαντήσω παραθέτοντας κάτι στα γαλλικά. Um, ίσως και να το πω και λάθος, αλλά τέλο πάντων περίπου λέει τα εξή. Δεν πρέπει ε, να ε, ελπίζουμε για να επιχειρήσουμε κάτι, ούτε και να περιμένουμε να πετύχουμε για να επιμένουμε στην προσπάθειά μας. Δηλαδή μπορούμε να τους μεταποιήσουμε ε, τους Κινέζους και βλέπετε το σχέδιο το πενταετές και το δεκαετές ότι έχει παίξει κάποιο ρόλο και είναι προς όφελος της ίδιας της Κίνας να επανισορροπηθεί το ισοζύγιο. Ε, το ποσοστό κατανάλωση στην Κίνα αντιστοιχεί στο 40% του ΕΠ. αυτό δεν είναι προ συμφέρον της ε, κινέζικης βιομηχανίας. Δεν έχουν κανένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας ε, πρέπει να αποταμιεύουν πολύ μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος ούτως ώστε να πάνε σε καλά σχολεία τα παιδιά του γιατί είναι πανάκριβη η φίτηση και δεν ε, υπάρχει παρά μόνο μια μηδαμινή ε, συνεισφορά από πλευρά του δημοσίου. Οι ίδιοι οι Κινέζοι δηλαδή πρέπει να φροντίσουν ούτως ώστε να αυξηθεί η ευμάρεια για όλους και ε, αργά αναδιαρθρώνουν, επαναπροσανατολίζουν ε, την κινέζικη αναπτυξιακή πορεία, αν θέλετε. Δεν το απάντησα αυτό το προηγουμένως, ε, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις, οποίες δεν πρέπει να απαντούμε. Μιλήσαμε για τη δημοκρατία στην Κίνα, μιλήσαμε για τον Ε, και μιλήσατε για το ρόλο της ε, G20 Φυσικά όταν συζητούμε με την Κίνα ε, ε, μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα και φυσικά όλα αυτά τα θέματα δημοκρατίας επηρεάζουν και την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον της Κίνας ε, και όταν λέτε ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και χάρη σε αυτό μπορούν ευκολότερα να λαμβάνουν αποφάσεις και να δρουν και ταχύτερα οι Κινέζοι θα σας έλεγα ότι οι δικοί μας για την Κίνα έχουν διαφορετική άποψη μας λένε πως ε, το σύστημα βασίζεται στη συνένεση σε τέτοιο βαθμό που πέρσι στο διάλογο ΕΕ Κίνας όταν φαινόταν ότι θα ήταν αδύνατο να καταλήξουμε σε συνένεση, ξέρετε τι ανάλυση έκαναν μεταγενέστερα, ότι έφτασαν, ε, έφτασε ο Πρωθυπουργό ε, της Κίνας στα όρια του. Δεν μπορούσε να τα υπερβεί, δεν μπορούσε να εγκρίνει άλλες συνενετικές λύσεις γιατί ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όταν μιλούσαμε για τις δικές μας συζητήσεις στο G20 και, λέμε, και έλεγα πριν στην πρώτη μου παρουσίαση ότι λένε όχι οι Κινέζοι και δεν συζητούν καν τα επιχειρήματά τους, είναι γιατί έχουν περιορισμούς, έχουν περιορισμούς εντελώ διαφορετικής ε, φύσεως και δεν μπορούν να δεχτούν κάποια πράγματα. Ε, Τώρα αυτά που ακούγονται ότι θα γίνουμε σαν την Κίνα, ότι θα εργαζόμαστε πολύ περισσότερες ώρες, θα πληρωνόμαστε λιγότερο, ότι οι Κινέζοι εργαζόμενοι θα έχουν τα, τις ίδιες παροχές και άρα δεν θα χρειάζεται να αποταμιεύουν τόσο πολύ και θα αυξηθεί η εγχώρια κατανάλωση. Όλα αυτά υπερβαίνουν το αντικείμενο του διαλόγου μας με τις κινέζικες αρχές. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Uh, Οι διαρθρωτικές τώρα αλλαγές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κίνα είπατε, ναι, αλλά νομίζω αναφερθήκατε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εκτεταμένα φαινόμενα που επηρεάζουν την ε, οικονομική ανάπτυξη της ε, Ένωσης. Δεν εννοούσατε αυτό. Κυρία Χιούπνερ, παρανόησα τότε την παρέμβασή σας. Um, Νόμιζα ότι με ρωτήσατε τις διαδικαστικές αλλαγές στην Ένωση. Λοιπόν, στην Κίνα. Μάλλον και εδώ πάλι θα σας πω δεν είμαι ο σωστός άνθρωπος για να σας απαντήσω. Παρ' όλα αυτά κατέχω τη θέση που κατέχω σήμερα. Όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζουμε στην Κίνα για να αιτιολογήσουμε τη θέση μας, τα περί διαρθρωτικών ε, αλλαγών, τα περί μεταρρύθμισης ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Λοιπόν, αυτός ο τομέας ε, κάνει επενδύσει όχι επί τη βάση των οικονομικών μεγεθών, αλλά σκέφτεται, α, πρέπει να γίνουν επενδύσει σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το τομέα, δεν ευελτιστοποιούνται όμω οι επενδύσει. Τέτοιου είδου διαρθρωτικέ αλλαγέ θα θέλαμε να εφαρμόσουν οι Κινέζοι και είπα προηγουμένω ότι θα πρέπει να μειώσουν την ε, μη αναδιανομή μερισμάτων, κυρίω στι δημόσιε επιχειρήσει, ε, γιατί υπάρχει πλημελή ε, κατανομή των πόρων στην Κίνα. Δηλαδή κάποιοι έχουν πελώρια κέρδη, δεν ξέρουν να τα κάνουν. Δεν μπορούν να δώσουν τα μερίσματα στους μετόχους γιατί δεν έχουν μετόχους, γιατί ο μόνος μέτοχος είναι το δημόσιο. Ε, ε, δηλαδή, από πολλές πλευρές δεν είναι βέλτιστες οι επενδύσεις ε, στην Κίνα και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν είναι άξια λόγου, αν θέλετε. By, by, αλλά Σίγουρα συμφωνούν όλοι ε, και λένε ότι οι πολλές αλλαγές θα ήταν όφελο τη Κίνα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει λοιπόν την πρώτη συζήτηση. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη, εάν ε, δεν έχετε άλλα ερωτήματα, αλλά θα κάνω και εγώ μια σύντομη παρατήρηση. Μου φαίνεται ότι στη συζήτηση αυτή ε, ότι φάνηκε ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό το ότι η Κίνα εξάγει τόσο πολύ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί προβλήματα, αλλά αυτό είναι μια αμερικάνικη απόφαση. Μια εταιρεία όπως η General Electric. Όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν απαιτούν υψηλή, πολύ υψηλή τεχνολογία, τα παίρνει από την Κίνα. Αυτό είναι μια αμερικάνικη απόφαση των αμερικανικών επιχειρήσεων. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την απόφαση του πολιτικού γραφείου του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος η Αμερική παίρνει σχεδόν τα πάντα και εισάγει σχεδόν τα πάντα από την Κίνα. Για τον κύριο Χουντή τώρα. Γιατί αναφέρθηκε στις ε, διαφορές που υπάρχουν ε, τις, τις ανισομέρειες μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε μια εσωτερική αγορά που δεν είναι απόλυτα συμπληρωμένη, αλλά Παρ' όλα αυτά, όταν έχουμε διαφορέ μεταξύ, μεταξύ Γερμανία από τη μια πλευρά και την Ελλάδα και την Πορτογαλία από την άλλη πλευρά, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα οποία εξάγει η Γερμανία κατά 55% εισάγονται από άλλε Ευρωπαϊκέ χώρε, όπω είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία κτλ. Δεν πάνε στην Αμερική. Κατά 55% τα προϊόντα αυτά πηγαίνουν σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Αν η Γερμανία εξάγει περισσότερο, τότε είναι επειδή εισάγουν λιγότερο αυτέ οι χώρε. Αν θέλει ο κόσμο να έχει γερμανικά αυτοκίνητα, παραδείγματο χάρη, εμεί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα εξαγάγουμε και να πάει ο κόσμο να αγοράζει πορτογαλέζικα αυτοκίνητα ή να παίρνει, ξέρω εγώ, κορνθιακέ σταφίδες. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Πρέπει να δούμε τα πράγματα λοιπόν πιο ρεαλιστικά. Μετά από αυτό το σχόλιο λοιπόν θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Συγγνώμη κύριε Μπίρξ, που θα σας ε, εκμεταλλευτούμε τόσο πολύ. Θα σας ε, δώσουμε και ένα καλό καφέ ίσως στο τέλος. Είναι κουραστικό κάπως για σας. Αλλά ξέρουμε ότι είσαστε προσιλωμένος να μας δώσετε τις απόψεις σας για το θέμα αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έρθουμε στο δεύτερο θέμα τώρα που είναι το νέο παγκόσμιο σύστημα ισοτιμιών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μα είναι ευχαρίστηση για μένα να είμαι μαζί σας και Χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον και ευφύης ερωτήσεις. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Έρχομαι λοιπόν στο δεύτερο θέμα, τη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία από τις προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας των G20 και η πρόσφατη ομιλία του Προέδρου Σαρκοζή για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στην ε, διπλωματική κοινότητα αναφέρθηκε στο σύστημα ισοτιμιών ως ένα μη σύστημα. Έτσι λέγαμε το 1976 την κατάσταση που επικρατούσε. Όπως και να το πείτε, το μη σύστημα ή εγώ θα έλεγα υβριδικό σύστημα, γιατί εμείς μιλάμε πια για ένα υβριδικό σύστημα, μας έχει εξυπηρετήσει σχετικά καλά τα τελευταία 40 χρόνια τόσο οι προηγμένες όσο και οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν περάσει μια μεγάλη περίοδο συνεχούς ανάπτυξης και σταθερών τιμών και η κρίση η χρηματοοικονομική του 2008 θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είχε να κάνει με κάποια αστοχία του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Το σύστημα ήταν αρκετά ανθεκτικό στην κρίση αυτή. Ζούμε λοιπόν στον βέλτιστο όλων των δυνατών κόσμων σε ένα κόσμο αγγελικό. Όχι. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Καταρχήν έχει αλλάξει ο κόσμος. Και η προηγούμενη μας συζήτηση το κατέδειξε αυτό. Η παγκόσμια οικονομία του 21ου αιώνα έδειξε ότι υπάρχει ανάδυση δύο σημαντικών παικτών στον οικονομικό στίβο. Μιλήσαμε για την Κίνα, αλλά υπάρχει και η Ινδία. Και όλα αυτά θα έχουν επίπτωση στο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Επίσης όμως είδαμε τα πρόσφατα χρόνια ότι το τωρινό σύστημα αντιμετωπίζει πάρα πολλές ατέλειες, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ποιες είναι λοιπόν οι δυσκολίες και οι ατέλειες. Καταρχήν, έλλειψη ευθυγράμμισης των ισοτιμιών. Όταν τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα της διακύμανσης των ισοτιμιών οι οικονομολόγοι, θεωρούν ότι η αστάθεια σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο των ισοτιμιών δεν οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα αλλά η οξία και συνεχιζόμενη έλλειψη ισορροπίας της ισοτιμίας μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα γιατί οδηγούν σε στρεβλώσεις <clears throat> σε ό,τι αφορά την αποταμίευση, την, ε, ε, τις επενδύσεις, την απασχόληση κτλ. Και αυτό το επιχείρημα έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές για τις ε, ισοτιμίες ε, Πολλές φορές όμως επανέρχονται στην κανονική τους τιμή οι ισοτιμίες. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με την ακαμψία των ε, ισοτιμιών, των σταθερών ισοτιμιών και εδώ φυσικά το καλύτερο παράδειγμα είναι η Κίνα. Η δεύτερη πηγή ανισομεριών είναι η αστάθεια των κεφαλοχικών ροών. Βλέπουμε πολύ μεγάλες ροές οι οποίες ακολουθούνται από απότομο σταμάτημα των ροών. Και φυσικά οι ροές κεφαλαίων θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες. Η ροή ας πούμε, κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές φαίνεται ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη γιατί τουλάχιστον εν μέρη αντανακλών, αντανακλούν μακροχρόνιες προοπτικές για καλή απόδοση στις ε, επενδύσεις και στα κεφάλαια. Η αστάθεια λοιπόν και οι διακυμάνσεις δεν είναι απόλυτα αρνητικές. Σε ορισμένε περιπτώσεις οι διακυμάνσεις, οι κινήσεις στις τιμές των, ανα, των στον τιμών των αγαθών των, του, στοιχείων του ενεργητικού βοηθούν το σύστημα να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Και αυτό ισχύει και για τα βασικά προϊόντα. Όλα αυτά κανονικά θα πρέπει να βοηθήσουν την παγκόσμια ευμάρεια διότι αντισταθμίζει την ακαμψία των βασικών προϊόντων. Η αστάθεια αυτή να γίνεται πρόβλημα βέβαια όταν δεν έχει να κάνει με ουσιώδεις λόγους και όταν οι χρηματοοικονομικές αγορές μπορούν να οξύνουν τους κλειδονισμούς και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μόνιμη αστάθεια η οποία δημιουργεί και κινδύνους για την πραγματική οικονομία. Μια τρίτη πηγή ε, αστάθειας έχει να κάνει με παγκόσμιες ανισομέρειες που συζητήσαμε και έλλειψη προσαρμογής απαραίτητης των πολιτικών. Εδώ είναι σφανερό ότι χρειάζεται να υπάρξει επανεξισορρόπηση της συνολικής ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί στους G20. Αλλά η συνεκτική στάση των G20 ούτως ή άλλως έχει μειωθεί εφόσον εξερχόμαστε από την χρηματοπιστωτική κρίτη. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι, ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες βασίζονται στο ότι ο καθένας θα τακτοποιήσει το σπίτι του και όλα πάνε καλά, αυτές είναι προβληματικές πολιτικές γιατί δεν είναι κακό να εξηγιάνει κανεί τα δικά του δημοσιονομικά και οικονομικά, αλλά πρέπει να δει και τον αντίκτυπο ο οποίο προκαλείται στου γείτονέ του από μια τέτοια πολιτική. Αν αυτέ οι πολιτικέ δεν τύχουν διεθνού συντονισμού και αν δεν λάβουν υπόψη το γεγονό ότι ξεπερνάει το αποτέλεσμα στην ίδια τη χώρα μια τέτοια πολιτική, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει λοιπόν από τις διαδικασίες αυτές τις μεμονωμένες τρόπος να αποφύγουμε τη δημιουργία ανισοτήτων και ανισομεριών και δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης αυτών των ανισομεριών. Αν υπάρχουν προσαρμογές πολλές φορές είναι ασυμμετρικές, μεγαλύτερη προσαρμογή γίνεται στις χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα και στις χώρες που δεν έχουν αποθεματικό νόμισμα από ότι στις υπόλοιπες χώρες οι οποίες έχουν δικό τους αποθεματικό νόμισμα. Ένα τέταρτο πρόβλημα είναι η διεθνής ρευστότητα και η συσσόρευση αποθεματικού. Αυτή τη στιγμή περίπου 60% των επισήμων συναλλαγματικών αποθεμάτων βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 60%, περίπου 30% σε ευρώ και 10% σε άλλα νομίσματα. Και στο διεθνές επίπεδο και στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές μόνο ένα μικρό φάσμα νομισμάτων χρησιμοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει κλειδό σε, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαδοθεί αμέσως και με μεγάλη ταχύτητα στον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ αν έχουμε μια κρίση σε άλλα μέρη του κόσμου τότε προσπαθεί κανείς να βρει ένα ασφαλές καταφύγιο και θα περάσει στα βασικά νομίσματα, όπως είναι το ευρώ ή το δολάριο. Αλλά η σταθερότητα του συστήματος σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξαρτηθεί απόλυτα από την σταθερότητα του πυρήνα, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν είναι ένα τέλειο σύστημα. Επομένως, το να βασιζόμαστε σε αυτούς οι οποίοι εκδίδουν τα νομίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε επίπεδο παγκόσμιο αποθεματικό, αυτό έχει δημιουργήσει αύξηση των ε, αποθεμάτων συναλλάγματος σε πολλές χώρες οι οποίες είναι αναδυόμενες. Η κάλυψη σε αυτές τις χώρες πολλές φορές είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό τους χωρέως. Αυτό είναι υπερβολικό να Το να σωρεύει κανεί τέτοιου πόρου, το να σωρεύει κανεί αποθεματικά δημιουργεί προβλήματα και σε επίπεδο κατανάλωση και σε επίπεδο επενδύσεων, γιατί υπάρχει ουσιαστικά μια, θα έλεγα, στασιμότητα στην κυκλοφορία των κεφαλαίων. Και για να σωρεύουν αποθεματικά, ορισμένες χώρες ακολουθούν πολιτικές ουσιαστικά προστατευτισμού επιδιώκουν θα έλεγα πλεονάσματα τα οποία πλεονάσματα στους τρέχοντες λογαριασμούς ε, οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή τη φάση. Το να προσπαθεί κανείς να βρει μια άκρη στην ε, υπόθεση αυτή μπορεί να το κάνει όταν ξεκαθαρίσει κάπως το, τις ευθύνες κάθε τμήματος και κάθε υπηρεσίας. Κάποιες πρώτες ιδέες βέβαια τις έχουμε και θα ήθελα να σας τις παρουσιάσω. Ξεκινώντας πάντα από τις διεθνείς αυτές ε, λήψεις ισορροπίας ή ανισότητες αν θέλετε. Θα πω κάτι που το έχω ήδη πει. Υπάρχει ανάγκη για μια αντιμετώπιση η οποία να εμπνέεται από πνεύμα συνεργασίας. Ε, καταρχάς σε επίπεδο ισοτιμιών. Εκεί απαιτείται να υπάρξει συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της συμφωνίας την οποία κατέληξαν στην ε, Σεούλ σε ένα σύστημα ισοτιμιών το οποίο να δείχνει ουσιαστικά το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό τμήμα της ανακοίνωσης της ΕΟΥΛ. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η βασική δυσκολία. Δεύτερον, θα πρέπει να βρούμε συνεχείς λύσεις, διαρκείς λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από τη σώρευση αποθεματικών και να δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των αποσταθεροποιητικών της κίνησης κεφαλαίων. Η σώρευση αποθεματικών αφεαυτής δεν είναι κάτι το, κακό ε, από μόνο του. Η Νορβηγία σαν παράδειγμα δημιούργησε ένα ταμείο από τα έσοδα ε, του πετρελαίου το οποίο έχει σαν προορισμό να βοηθήσει τον πληθυσμό. Αυτό δεν είναι κακό αλλά εκεί όπου δημιουργείται κάτι το κακό είναι όταν υπάρχει υπερβολική σώρευση. Και τι γίνεται όταν προσπαθεί κανείς να, να αποτρέψει μια τέτοια υπερβολική σώρευση. Ίσως πρέπει να βοηθηθούν ορισμένες χώρες να κατανοήσουν ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο αποθεμάτων. Δεν είναι εύκολο να το γνωρίζουν οι χώρες αυτές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρούμε ότι η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική και ελπίζουμε να καταλήξει στο να βοηθήσει ε, τις χώρες οι οποίες έχουν το πρόβλημα αυτό. Το θέμα δεν είναι αρκεί εκεί βέβαια, δεν περιορίζεται εκεί. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ουσιαστικές αιτίες της όρευση αυτής. Τις περισσότερες περιπτώσεις είναι η ανάγκη για μια αίσθηση ασφάλειας. Θυμηθείτε λίγο την Ασία. Οι ασιατικές χώρες έχουν περάσει προβλήματα σοβαρά στην ασιατική οικονομική κρίση του 1997-98. Τότε ήταν κρίση αποθεμάτων. Εκεί ακριβώς αυτή η έννοια της ασφαλείας ήταν καθοριστική. Πώς μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Μπορούμε να παρέχουμε σαν παράδειγμα εναλλακτικά δίκτυα ασφαλείας οικονομικά για χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν έλλειψη διεθνούς ρευστότητας. Στα πλαίσια της ομάδας των 20 έχει επιτελεστεί αρκετά σημαντική πρόοδος. The financial instruments. More still needs to be done in order to... έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε δίκτυα ασφαλείας, εξετάζουμε τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους From Πώς τα χρηματοπιστωτικά σοκ, σαν παράδειγμα, μεταδίδονται από τη μία χώρα στην άλλη. Λοιπόν, πώς μπορούμε να παρεμποδίσουμε δηλαδή μια διάδοση ενός φαινομένου αρνητικού όταν αρχίζει αυτό να εκφράζεται. Πώς μπορούμε επίσης να διαμορφώσουμε περιφερειακά δίκτυα ασφαλείας, τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο περιφερειακό σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε ότι υπάρχουν και στην Νοτιοανατολική Ασία κάποια τέτοια δίκτυα και θα πρέπει όλα αυτά να συντονιστούν με τα προγράμματα του ΔΕΛΤΑ και επίσης ε, θα πρέπει οι εμπειρίες μας να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης με την καλή έννοια από άλλες χώρες και στον τομέα ε, της αιρεσιμότητας και στον τομέα των προϋποθέσεων μάλλον και σε άλλους τομείς. Μια άλλη ιδέα η οποία είναι υπό εξέταση, κυκλοφορεί ε, είναι το πέρασμα σε ένα πολυπολικό σε εισαγωγικά σύστημα αποθεματικών. Έτσι θα μειώσουμε την έκθεση των συστημάτων σε κινδύνους οι οποίες να προέρχονται από μεμονωμένες χώρες, όπως στο παρελθόν πρόσφατα από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πιστεύουμε ότι οι διακυβερνήσεις, οι οικονομικές και οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να δημιουργήσουν την δυνατότητα αποθεματικών με πολλούς τρόπους, όχι δηλαδή μονομερείς οι χώρες θα αποφασίζουν αν θα αγοράζουν ένα νόμισμα ή δεν θα αγοράζουν αυτό το νόμισμα έτσι ώστε ένα συγκεκριμένο νόμισμα να μην είναι καθοριστικό απόλυτα για μια οικονομία και ανάλογα με την τύχη που θα έχει το νόμισμα αυτό να επηρεάζει μια οικονομία ε, περισσότερο από όσο θα έπρεπε, από όσο είναι ε, φυσιολογικό. Νομίζω επίσης ότι αυτό είναι κάτι που έχει άμεση σχέση με το βάθος και τη ρευστότητα των αγορών που εργάζονται κυρίως από το αμερικανικό δολάριο γύρω. Θα πρέπει να δώσουμε επίσης και στα SDR, δηλαδή ε, στις δυνατότητες τις οποίες έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το προσωπικό του Δέλτα Νιτάφ προετοίμασε ένα έγγραφο πρόσφατα και αυτό το οποίο προτείνουν είναι καταρχάς τα SDR να αποκτήσουν ουσία. Αυτά τα δικαιώματα έκδοσης του ΔΝΤ θα πρέπει να ευξηθούν επίσης πάρα πολύ αυτά τα δικαιώματα έκδοσης γιατί προς στιγμή η ποσοτική τους παρουσία είναι ελαχιστότατη σε σχέση με τα αποθέματα τα οποία υπάρχουν. Για να μπορέσουν τα SDR να καταστούν χρήσιμα τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα απαιτείται να υπάρξουν ορισμένες νομικές αλλαγές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πλήρως. Εμείς την πρόταση αυτή την έχουμε σε μια φάση εξέτασης σε αυτή τη φάση. Δεν έχουμε εκφραστεί για το αν είναι μια θετική ε, πρόταση ή μια πρόταση που παρουσιάζει προβλήματα. Αυτά τα ειδικά εκδοτικά δικαιώματα ή τραβηκτικά δικαιώματα. This brings me Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος ε, προηγουμένως αναφέρθηκε σε ένα άλλο θέμα για το αν θα πρέπει να διευρύνουμε το καλάθι του SDR για να συμπεριλάβει και το κινέζικο νόμισμα. Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο την ενίσχυση του ίδιου του ρόλου των SDR, αυτών των δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα έτσι θα καταστήσουμε το κοινωνικό νόμισμα ένα νόμισμα το οποίο να λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν επίσης και προβλήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε στην Κίνα ιδιαίτερα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, άνοιγμα κεφαλαιοχικών αγορών να υπάρξει ένα ουσιαστικό, ε, ε, μια ουσιαστική κεντρική ανεξάρτητη τράπεζα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν στην Κίνα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις αποσταθεροποιητικές τάσεις των κεφαλαιοκικών ροών. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη ομοβροντία θα έλεγα εποπτείας και ελέγχου των κεφαλαιοχικών χωρών από πάρα πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και από τις χώρες της ομάδας των 20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το φαινόμενο είναι ασυχητικό. Θεωρούμε ότι το ελεύθερο, η ελεύθερη κυκλοφορία των οικονομιών είναι ευεργετική για την οικονομία. Και αυτό περιλαμβάνεται επίσης και ε, στις συνθήκες. Απαγορεύεται ο έλεγχος ε, το, του κεφαλαίου. Όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ανάμεσα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος της κυκλοφορίας του κεφαλαίου λοιπόν δεν είναι η καλύτερη λύση όταν συγκριθεί με κάποιες άλλες λύσεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι καλύτερες, όπως κάποιες πολιτικές μακροοικονομικής σταθερότητας, όπως επίσης και κάποιες ε, πολιτικές λογιστικού ελέγχου, οι οποίες να λειτουργούν μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικά. Απαιτείται λοιπόν αυτές οι σταθεροποιητικές πολιτικές να περιορίσουν γενικά τους κύκλους ε, υπερβολικής αύξησης μιας οικονομικής δραστηριότητας που διαδέχεται ένας άλλος κύκλος ε, μείωσης κτλ. Βλέπουμε ότι αυτές οι βίες αλλαγές είναι αρνητικές. Η επιρροή αυτών των κινήσεων είναι πάρα πολύ ισχυρή και σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος των κεφαλαιαγορών θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση. Είναι η τελευταία λύση, θα πρέπει να είναι κάτι το προσωρινό θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονική διάσταση, θα πρέπει να είναι ειδικά στοχευμένη, όχι γενικά όλες οι αλλαγές, όλες οι κυκλοφορίες και οι ροές. Και δεύτερον θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο συντονισμού σε πολυμερές επίπεδο. Είναι αρνητικό για τη διεθνή συνεργασία ορισμένες χώρες να εισάγουν αυτού του τύπου την εποπτεία και τους ελέγχους και να παρεμβαίνουν στις αγορές των ισοτιμιών χωρίς να έρχονται σε διαβούλευση με τις υπόλοιπες χώρες, με τους εταίρους τους. Συνεπώς λοιπόν οι έλεγχοι αυτοί δικαιολογούνται μόνο σε περιπτώσεις χωρών οι οποίες έχουν υπερτιμημένα ε, επίπεδα ισοτιμιών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι θεωρητικά υπεύθυνο για αυτές τις ε, ε, κινήσεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα σημαντικός ρόλος για το ΔΝΤ στις ροές αυτές και είμαστε υπέρ του να υπάρξει μια ξεκάθαρη εντολή προς το Δέλτα Νιτάφ για την χρήση αυτών των μορφών ελέγχου. Όπως προτάθηκε πρόσφατα και από την κυρία Λαγκάρντ Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέρ για την πλήρη σας παρουσίαση και εισαγωγή στο δεύτερο μέρος. Έχουμε τώρα μία σειρά από ομιλητές οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο η Περβάνς και ο Σάνσες Πρεσέδο, μετά ο Γκέμπελς και ο Όλε Σμιτ, ο Μιγγέλ Πόρτας και ο κύριος Κυλακάκης. Αυτά προς το παρόν. Η εισηγήτριά μας η Περβάνς Μπέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση. Έχω μία πρώτη κάπως χαζή ερώτηση. Για την επόμενη συνάντηση ε, του G20 υπάρχουν ισχυρές ε, φιλοδοξίες ε, και μεταξύ των θεμάτων είναι και η αναδιοργάνωση του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Με ποια κριτήρια θα εκτιμ θα κρίνατε εσείς ότι είναι χρήσιμο το G20. Τι μπορούν να περιμένουν οι Ευρωπαίοι από τη συνεδρία της ομάδας G20. Δεν πρόκειται φυσικά εμείς να αμφισβητήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ταυτόχρονα βέβαια διαπιστώνουμε ότι στο carry trade ε, αυτή η κυκλοφορία των κεφαλαίων μπορεί να οδηγήσει σε κερδοσκοπικές ε, ε, κινήσεις και ζητείτε μετά προσπάθεια από τους λαούς της Ευρώπης για να περάσουν τα ε, διαρθρωτικά προγράμματα. Κάποιοι τα ονομάζουν διαρθρωτικά προγράμματα, άλλοι τα ονομάζουν τις προσπάθειες πολιτικές λιτότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να υποστηρίξει τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρώτον και δεύτερον προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια ε, σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος ε, μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ νομισμάτων, αυτό το διάσημο carry trade. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω και εγώ μερικά ερωτήματα. Καταρχήν, η Γαλλική Προεδρία στους G20 έχει το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη προφανώ. Τι είδου συντονισμό υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ του Προέδρου τη Ευρωομάδο, τη Κομισιόν και της Γαλλικής Προεδρίας των G20 για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Δεύτερον, ένα ερώτημα μακροοικονομικού χαρακτήρα. Λέτε ότι το νομισματικό σύστημα επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά μας. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, αλλά αν ανεβαίνει η ισοτιμία του νομίσματός μας, όλες αυτές οι προσπάθειες πέφτουν στο νερό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το δολάριο να υποτιμάται και μαζί του οι τιμές των βασικών προϊόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένως πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που κάνουμε επηρεάζονται από όλα αυτά. Και εξάλλου το νομισματικό σύστημα έχει να αντιμετωπίσει πολλούς ε, στόχους. Δεν μπορούμε αυτό να προσπαθήσουμε να το κάνουμε με πολυετή στόχους και με μια κοινή συνένεση. Να έχουμε μια μακροοικονομική συνεργασία όπως είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Το σύστημα του Bretton Woods χρησιμοποιούσε βασικά στοιχεία τα οποία ήταν ουσιαστικά μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες. Το σύστημα του GATT, το οποίο ήταν παιδί του Bretton Woods. Δεν υπάρχει πια το σύστημα του Bretton Woods, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το βασικό στοιχείο το οποίο απαρτίζουν οι κινήσεις κεφαλαίων. Έχουμε ένα πολυμερές σύστημα για το παγκόσμιο εμπόριο. Μήπως πρέπει να υπάρχει και ένα πολυμερέ σύστημα για τι κινήσει κεφαλαίων. Όλοι θέλουμε να υπάρχει ελευθερία κίνηση κεφαλαίων, αλλά θέλουμε να έχουμε σταθερότητα και αηφόρο ανάπτυξη. Μήπω είναι λοιπόν απαραίτητο να εξασφαλίσουμε κάποια ισορροπία και για τι κινήσει κεφαλαίων. Όταν πήγαμε στην Ινδία και συζητήσαμε με τι Ινδικέ Αρχέ, αυτά τα οποία ακούσαμε έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στι χώρε αυτέ από τι μεγάλε εισρωέ κεφαλαίου πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν ε, στη δεκαετία του 90 στο Μεξικό, στις ασιατικές χώρες, στην Τουρκία, όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα μεγάλων κερδοσκοπικών εισρώων κεφαλαίων που στη συνέχεια έφυγαν. Λοιπόν, η είσοδοι κεφαλαίου, όταν θέλουμε να γίνουν επενδύσεις, είναι καλό αυτό το πράγμα. Αλλά όταν δεν έχουν τέτοιο χαρακτήρα, οι εισρώες κεφαλαίου θα πρέπει να υπόκειται σε κάποιες ε, σε κάποιε μορφέ ελέγχου. Αν μπαίνουν σε μια χώρα, δημιουργούν μια κατάσταση ανεξέλεγκτη και μετά η χώρα πρέπει να κάνει προσαρμογέ, αυτό δεν είναι θετικό. Μήπω πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα πολυμερέ σύστημα για να ελέγχουμε τι ροέ κεφαλαίων και να εξασφαλίσουμε ότι οι αγορέ ε, αξιογράφων δεν θα έχουν απότομε διακυμάνσει και ότι οι αγορέ των ε, αμερικανικών αξιογράφων χρηματο, μπορούν να έχουν ένα σταθερό χαρακτήρα για να αντιμετωπίσουν τις χώρες αυτές. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν μια παγκόσμια ρύθμιση του εμπορίου χωρίς να υπάρχει και αντίστοιχη ρύθμιση στον τομέα των χρηματοοικονομικών. Μήπως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πράγμα. Επίσης στα θέματα των ισοτιμιών. Είναι σαφέ ότι πρέπει να υπάρξει κάποια προσαρμογή στι συνθήκε αγορά και να υπάρξει και κάποια ανταγωνιστικότητα. Και οι βασικέ οικονομίε θα πρέπει να φέρουν τα νομίσματά του σε ένα κοινό καλάθι. Όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Και ένα τελικό στοιχείο. Όλα αυτά τα θέματα που γίνονται σε νομισματικό επίπεδο απαιτούν μια νέα συμφωνία Bretton Woods. Η τελευταία συμφωνία του Bretton Woods έγινε το 1944. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινό. Μήπω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο όπω αυτό των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε ένα Συμβούλιο Ασφαλεία για τα πολιτικά θέματα. Μήπω πρέπει να έχουμε ένα Συμβούλιο Ασφαλεία για τα οικονομικά θέματα, ώστε και το σύστημα του διεθνού Νομισματικού Ταμείου που είναι προηγούμενο από τη δημιουργία του ΟΗΕ να μπει και αυτό σε αυτό το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Όπως είπα και στην αρχή, ε, είμαστε σε αρχικό στάδιο προβληματισμού για όλα αυτά τα θέματα. Το ίδιο σε σχέση με τον προβληματισμό που έχουμε για τις παγκόσμιες ανισομέρειες που ζητούσαμε προηγουμένως. Ε, έχω κάποιες απαντήσεις, αλλά κάποια ζητήματα ακόμη δεν έχουν αναλυθεί, κυρίως αυτό του carry trade ε, των μεταφορών κεφαλαίων μεταξύ νομισμάτων. Τουλάχιστον ε, δεν γνωρίζω εγώ να έχει γίνει κάποια ανάλυση της έννοιας του carry trade. Μας είπατε στο τελικά πώς θα κρίνουμε τα αποτελέσματα του G20, αν ήταν επιτυχής η συνεδρίαση ή όχι. Ε, ε, κοιτάξτε, για να είμαι και λίγο σοβαρός, θα έλεγα ότι θα χρησιμοποιήσουμε ως γνώμονες πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Και αυτό συνδέεται με την ερώτηση του κυρίου Σάντσες. Πώς θα γίνει ο συντονισμός με την προεδρία του Eurogroup κτλ. Κοιτάξτε, σε τεχνικό επίπεδο το συζητήσαμε αυτό το θέμα και σε άτυπο εξάλλου με την ε, Γαλλική Προεδρία στο παρελθόν. Η Γαλλική Προεδρία του G20 δεν έχει κάποιο μεγαλεπίβολο σχέδιο που φιλοδοξεί να επιβάλλει σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει πολύ συγκεκριμένε ιδέε σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του Διεθνού Νομισματικού Συστήματο. Ε, δεν είναι αυτή η στάση του. Θέλουν να ακούσουν τι απόψει όλων να τις αναλύσουν ε, ούτως ώστε να βελτιωθεί το σύστημα. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για επανάσταση. Θα τροποποιηθεί ένα υπάρχον σύστημα. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, υπάρχουν και επιμέρους ε, στοιχεία που μπορούμε να συζητήσουμε. Παραδείγματο χάρη τα κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Χρειαζόμαστε ασφαλιστικούς μηχανισμούς, κυρίως για τις ε, χώρες που γνώρισαν ε, τις ελλείψεις, σοβαρές ελλείψεις στα αποθεματικά τους ε, και πλήγησαν από αυτό τα περασμένα χρόνια και επίσης χώρες που αναγκάστηκαν να αναλάβουν ε, μέτρα αφού τους το ζήτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, παραδείγματος χάρη, έχουν τραυματιστεί σοβαρά από αυτό. Ε, και ε, δεν εννοούν να αποσυσσωρεύσουν τα αποθεματικά τους αν θέλετε. Τώρα, ε, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί για να μειωθούν τα αποθεματικά αυτών των χωρών και αν λειτουργούσε ένας τέτοιος μηχανισμός θα είχαμε και συγκεκριμένη πρόοδο. Για τα SDR τώρα, τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα. Δεν βάλουμε αμέσως το κινέζικο νόμισμα μέσα στο καλάθι των νομισμάτων, αλλά υπάρχει η ιδέα να διευρύνουμε, αν θέλετε, το περιεχόμενο του καλαθιού, κατόπιν συμφωνίας όλων των ενδιαφερομένων. Δεν μπορώ τώρα να επινοήσω συγκεκριμένα βήματα για τη μεταρρύθμιση των ειδικών τραβηχτικών δικαιώματων τώρα, αυτή τη στιγμή, αλλά πάντως για ε, τον χρηματοπιστωτικό κανονισμό και παρακολούθηση δεν είμαι ειδικό, αλλά ε, πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις γιατί θα τεθούν πολλά ζητήματα φέτος και πραγματικά αναμένονται από διάφορες πλευρές ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για τον ειδικό φόρο επιχρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, μιλήσατε για την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, του 2010. Εκεί λοιπόν ε, υποστηρίζει το φόρο ε, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, ανέλαβε τη δέσμευση να διερευνήσει περαιτέρω την εκπόνηση αυτού του φόρου επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, FTT όπως είναι γνωστό, σε συνεργασία με τους σημαντικότερους παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί ότι είναι κατάλληλο αυτό το εργαλείο του φόρου γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της ε, ε, επανακατανομής, της λανθασμένης ε, ανακατανομής των πόρων και θεωρούμε ότι σε παγκόσμιο και άρα διαρροής κεφαλαίων και άρα πιστεύουμε ότι υπάρχουν πλέον ενδεδειγμένα μέτρα, άλλα πιο ενδεδειγμένα μέτρα που μπορούμε να αναλάβουμε. Το θέμα στην, στο G20 είναι ότι οι εταίροι μας, όπως ε, οι Αμερικανοί, ούτε θέλουν να ακούσουν ε, τα περί FTT και όχι μόνο να συμμετάσχουν, όχι, ούτε καν φυσικά να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο σύστημα. Και αυτή είναι η βασική δυσκολία του φόρου αυτού. Σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι για να ισχύει σε ένα τέτοιο σύστημα. Τα περί συντονισμού τα σχολίασαν νωρίτερα και άτυπα αλλά και στην ομάδα εργασία του Eurogroup για τα οικονομικά και νομισματικά ζητήματα. Τα έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα γιατί εκεί επεξεργαστήκαμε και αυτά τα terms of reference, του όρου τη συμφωνίας που σας έλεγα. Κάτι ενσυχητικό βέβαια είναι ο εξής κίνδυνος. Ε, το άθος αυτό της προσαρμογής ε, ε, θα το επομιστεί σε πολύ μεγάλο κομμάτι η ζώνη ευρώ, δυστυχώς. Ε, εάν υπάρξει υποτίμηση δολαρίου, ε, οξυνθούν και άλλο οι ανισορροπίες. Ε, συνεχίζει να είναι υποτιμημένο και το ε, τότε όντω θα είναι ε, ε, ανησυχητικέ αυτέ οι τάσει και θα δημιουργηθούν βασικά ε, χρηματοοικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη. Εμεί προφανώς θέλουμε να το, να το αποφύγουμε και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ασκούμε πίεση στους εταίρους μας, όχι μόνο στην Κίνα, ούτω να είναι πιο διαλλακτική, αλλά ε, πιέζουμε και τις ΕΙΠΑ γιατί το έλλειμμά του υπερβαίνει το 10%. Πρέπει να εξηγιανθούν δημοσιονομικά και οι Αμερικανοί, ε, διότι ελοχεύει ένα σοβαρότατο κίνδυνος, ε, πιστεύουμε εμείς για τον παραλληλισμό που κάνατε με τον ΚΑΤ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπόριου και το, τα ή έναν αντίστοιχο διεθνή οργανισμό που θα μπορούσε να διαχειρίζεται τις κεφαλαιακές ροές. Ναι, αυτό είχα κατά νου στην πρώτη μου εισήγηση όταν σας είπα ότι θα μπορούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λάβει αυτό το χρήσιμο ρόλο και να εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των κεφαλαιακών ροών, τον, ε, την παρακολούθηση αυτών των ροών και το, κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένα καταξιωμένος οργανισμός ε, και μέσα ε, στην εντολή του προβλέπεται ο έλεγχος ε, το, του, χρηματοπιστωτικού συστήματος και άρα κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσε να αναλάβει και τον έλεγχο των κεφαλαιακών ροών. Είναι ο πλέον ενδεδειγμένος διεθνής οργανισμός για να αναλάβει αυτό το ρόλο, εν πάση περιπτώσει. Σχετικά τώρα με αυτά που είπατε για ένα ευρύτερο σύστημα, ε, ε, μιλήσατε για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τι να σας πω. Ε, και πάλι εδώ επανερχόμαστε στα ίδια. Δηλαδή, ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και στην αντιπροσωπευτικότητα. Τηρουμένων των αναλογιών θα μπορούσε κάποιο να θεωρήσει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο G20 και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ε, και ποια θα ήταν η γενική συνέλευση δηλαδή του ΟΗΕ, ποιο θα ήταν το αντίστοιχό της. Είναι δεν ξέρω, αυτά που είπατε για έναν ε, μεγάλο διεθνή οργανισμό που θα μπορούσε να συζητά αυτά τα προβλήματα, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η μέθοδο. Ρόμπερτ Γκέμπελς και Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μάθω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπόψη της κάποιες εξελίξεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών σε 50 πολιτείες και σε μεγάλες πόλεις. Όλοι γνωρίζουν ότι τα σφαιρικά ελλείμματα, το ομοσπονδιακό έλλειμμα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ζώνης ευρώ και δεν αναφέρομαι στην Ιαπωνία ή σε κάποιες άλλες χώρες. 48 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ελληματικούς προϋπολογισμούς και πολλές φορές εξαιρετικά ελληματικούς όπως το Ιλινόι, η Καλιφόρνια Καλιφόρνια έχει ένα θα έλεγα δημοσιονομικό χάσμα 50% περίπου. Λοιπόν, τι γίνεται με τα λεγόμενα δημοτικά ομόλογα, τα municipal bonds, τα οποία εκδίδονται είτε από τις μεγάλες πόλεις είτε από τις πολιτείες στη ΣΥΠΑ. Υπάρχει επίσης μια σχετική αύξηση ε, των επιτοκίων, ένα είδος ε, θα έλεγα πριν ε, κινδύνου το οποίο καλούνται να πληρώσουν αυτοί που τα αγοράζουν και ταυτόχρονα από ό,τι διαβάζω οι αγορές είναι θα έλεγα σε ακινησία πλέον. Οι επενδυτές δεν θέλουν να αγοράζουν αυτά τα ομόλογα. Πώς κρίνεται λοιπόν αυτό το τεράστιο χρέος που έχουν εσωτερικά οι ΙΠΑ και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές ή η κατάσταση στο εσωτερικό των ΙΠΑ. Όλε Σμιτ, η πρώτη ερώτησή μου έχει και αυτή σχέση με το δολάριο. Για πείτε μου, γιατί το δολάριο παραμένει το νόμισμα το οποίο εμπιστευόμεθα. Όχι μόνο Θεός το εμπιστεύεται όπως λέει, αλλά και εμείς. Αν ε, επισκεφθεί κανείς αφρικανικές χώρες με στενούς δεσμούς με την Ευρώπη, το δολάριο ε, πρέπει να χρησιμοποιήσει για να πληρώσει το ταξί του. Είναι θέμα εμπιστοσύνης μόνο και αν είναι θέμα εμπιστοσύνης είναι τόσο ανέφικτο να αλλάξει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη που μπορεί να εμπνεύσει. Έχουμε αρκετά προβλήματα και μέσα σε αυτά τα προβλήματα νομίζω τα προβλήματα αυτά είναι τόσο σοβαρά που μπορούμε πλέον να μιλάμε για αλλαγές. Δηλαδή το σύστημα λειτουργεί κάτω από τις παρούσες συνθήκες με αποτελεσματικό τρόπο. Όταν λέτε ότι θέλετε ένα πλήρως ανταλλάξιμο ρεμίμπι στην Κίνα και μία ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, έρχομαι στην προηγούμενη συνάντηση. Η δημοκρατία πού είναι. Γιατί δεν λέτε ότι η Κίνα χρειάζεται δημοκρατία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συζητάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά ε, θα ήθελα να μείνω σε αυτές τις ερωτήσεις για το δολάριο και για το ρεμίνμπι. Ε, στην ουσία εδώ βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια σφίκα. Η σφίκα ουσιαστικά επιστημονικά δεν πετάει. Δεν έχει τη δυνατότητα να πετάξει η σφίκα. Αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνει. Το ίδιο ισχύει και με την ερώτηση του Γκέμπελς θα έπρεπε ουσιαστικά όλε αυτέ οι πολιτείε να έχουν πτωχεύσει. Παρ' όλα αυτά δουλεύουν και παρ' όλα αυτά και εμεί αγοράζουμε δολάρια. Γιατί. Okay, good. Then go ahead. Yes. Παρακαλώ, ναι. Ίσως θα είναι πιο εύκολο να υπάρξει συνολική απάντηση. όλα αυτά που λέμε από τους εμπειρογνώμονες και από αυτά που λέτε κι εσείς ο ίδιος, φαίνεται ότι τώρα είναι η στιγμή που αναδύεται αυτό το νέο νομισματικό σύστημα και βλέπω να υπάρχουν πολλά δείγματα, πολλά σήματα του γεγονότος ότι προχωρούμε προς ένα σύστημα με πολλαπλά διεθνή νομίσματα. Το ερώτημά μου σχετίζεται με το εξή. Είπατε ότι έχουμε τώρα μια ανισομέρεια στην ανάπτυξη, ανισότητες, όλα αυτά μας υποχρεώνουν να δράσουμε, αλλά οι δράσει μα δεν είναι συντονισμένε αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν πολλέ σημαντικέ οικονομίε, όχι μόνο η Κίνα, που ακολουθούν ε, πολιτικέ δικέ του για το δικό του νόμισμα, που οδηγούν σε μεγάλε εντάσει στι παγκόσμιε αγορέ νομισμάτων. Υπάρχει το πρόβλημα το, ε, τον, τον στις κεφαλαίου <clears throat> ότι δεν υπάρχει φορολογία στι χρηματοοικονομικέ συναλλαγέ ότι θεωρούν ω ultima ratio οι περισσότερε χώρε το να εμποδίσουν τι ροέ κεφαλαίου και κάποια νομίσματα όπω το ευρώ είναι σίγουρα υπερτιμημένα. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση που δεν βρισκόμαστε σε σημείο ισορροπία, είμαστε μάλλον εκτό ισορροπία. υπάρχουν πολλέ στρεβλώσει στι αγορέ. και δεν έχουν προσαρμοστεί τεχνικά πλαίσια. Όταν αναδύονται λοιπόν όλα αυτά, τι είδου σύστημα θα μπορούσε να προκύψει από αυτές τις καταστάσεις όταν έχουμε τόσο μεγάλο υπόβαθρο στρεβλώσεων ή διαδικασιών που δεν τις καταλαβαίνουμε και που θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες σταθεροποίησης για να δημιουργήσουμε ένα νέο σταθερό πλαίσιο. Και το ερώτημα μου είναι, μπορεί ένα υγιές σύστημα το οποίο θα εκπληρεί τα κριτήρια τα οποία εσείς αναφέρατε να εξέλθει από αυτό το μπάχαλο. Μπορεί να βγει κάτι τέτοιο από την τωρινή κατάσταση. Ή μήπως πρέπει αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ή πρέπει να ξεπεράσουμε λύσεις οι οποίες ήταν απλώς εμβαλωματικές και προσωρινές. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε και να εδραιώσουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε όταν είναι μια κατάσταση τόσο ρευστή σε σχέση με τις αγορές και τις πολιτικές. Ευχαριστώ. Πρωτού αντιμετωπίσω αυτό το θέμα, που είναι πολύ θεμελιώδης ερώτημα, θα περάσω σε ένα θεμελιώδες και εξίσου ζωτικό πρόβλημα που είναι το θέμα των ελλημάτων των πολιτιών στις Ηνωμένε Πολιτείε και επίσης και κομιτιών και δήμων και κοινοτήτων στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι, η Κομισιόν εξετάζει το θέμα αυτό και αυτό είναι τμήμα της ανησυχίας που αντιμετωπίζουμε όταν μιλάμε με τους Αμερικανούς φίλους μας όταν εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τα δημοσιονομικά ελλείμματα των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριλαμβάνονται και οι πολιτείες και οι κομιτείες και οι δήμοι και οι κοινότητες. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι τμήμα του ελλείμματος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης αλλά είναι πρόσθετα στοιχεία τα οποία επιδεινώνουν το πρόβλημα. Τούτου λεχθέντος δεν είναι πολλά περισσότερα που μπορούμε να πράξουμε ως Κομισιόν παρά μόνο να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας προς τους εταίρους μας. Αλλά αυτό συνδέεται με το γεγονός του γιατί το δολάριο είναι ακόμα το κύριο διεθνές νόμισμα. Υπάρχει μια τεράστια ε, αδράνεια σε σχέση με το νομισματικό σύστημα. Είδαμε ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μάλλον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το αμερικανικό νόμισμα υπερκέρασε όλα τα άλλα όπως και τη Στερλίνα διότι η οικονομία των ΗΠΑ είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη ευρωστία έναντι της Αγγλικής ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είδαμε λοιπόν αυτή την κατάσταση σε σχέση με το ευρώ το οποίο υπάρχει μόνο εδώ και 11 χρόνια ουσιαστικά. Έχει κερδίσει κάποιο μερίδιο αγοράς αλλά δεν είναι το ίδιο μερίδιο αγοράς ε, όπως του δολαρίου και δεν έχει το ειδικό βάρος του δολαρίου στην παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει η αδράνεια, υπάρχουν τα φαινόμενα διαδικτύωσης. Αν κάποιος χρησιμοποιεί το δολάριο και εσείς χρησιμοποιείτε το δολάριο κατά ανάγκη, υπάρχουν πολλά σημαντικά ψυχολογικά προβλήματα Λέμε ότι οι άνθρωποι πάντα θεωρούν ως ασφαλές καταφύγιο το δολάριο, από τα γενοφάσκια τους θεωρούν το δολάριο είναι ασφαλές, οπότε το κάνουν και τώρα όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Είναι όπως παλιά αγόραζε ο κόσμος χρυσάφι. Τώρα τι νόημα έχει να αγοράσει κανείς χρυσάφι. Επομένως δεν μπορώ να σας δώσω περαιτέρω εξηγήσει στα φαινόμενα αυτά. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι ο ρόλος του αμερικανικού δολαρίου θα μειωθεί, γιατί ούτως ή άλλως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι η πιο σημαντική οικονομία σε παγκόσμιο κόπο. Ο κύριος Γκούμπελς, αν μπορώ να παρέμβω εδώ, είχα πάει να ακούσω μία διάλεξη από ένα καθηγητή από το Μόναχο, που είπε ότι είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο το δολάριο έχει δεσπόζουσα θέση γιατί οι κεφαλαιαγορές κυριαρχούνται από αγγλοσάξονες τραπεζίτες και προσπαθούν αυτοί να επιβάλλουν την άποψή τους. Uh, Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να μιλήσω κατά αυτόν που λέει ο Τσιν. Νομίζω όμως η μεγαλύτερη αγορά είναι το Λονδίνο στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη δηλαδή έχουμε Αγγλοσάξονες. Η υποψία μου λοιπόν για την εξήγηση αυτή και για να υπάρξει μια, ένα οικονομικό όφελος για την εγκατάλειψη αν θέλετε του, του δολαρίου προς ε, το Ζιμπαμπουενό δολάριο. Αν υπήρχε βεβαιότητα για οικονομικό κέρδος θα το κάναμε. Σχόλια χωρίς μικρόφωνο από την αίθουσα. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα εδώ παραμένει χένον και για τον κύριο Τζιν. Κάτι το οποίο μας παρηγορεί. Άμα δεν ξέρει αυτός, πώς να ξέρουμε εμείς. Σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Χιούμπνερ. Αυτό το οποίο προσπάθησα να πω είναι ούτε εμεί ούτε καν ο κύριο Σαρκοζή δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μαγικό μα καπέλο ένα νέο σύστημα. Το θέμα είναι να έχουμε ένα σύστημα στη διάθεσή μας το οποίο έχει δουλέψει καλά τα τελευταία 40 χρόνια και δεν καταστράφηκε από την οικονομική κρίση. Μπορεί να μην έλυσε εντελώ την οικονομική κρίση αλλά δεν προκάλεσε το ίδιο την οικονομική κρίση. Α μην πετάξουμε το μωρό λοιπόν με το νερό μαζί Ας προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις αδυναμίες τις οποίες έχουμε. Είπα ότι έχουμε αδυναμίες στον τομέα των ισοτιμιών, στον τομέα των ορών, των κεφαλαίων. Έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Ας προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε, βρίσκοντας τρόπους σαν παράδειγμα παροχής διεθνούς ρευστότητας η οποία να μην προέρχεται υποχρεωτικά από την κεντρική χώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη ΣΥΠΑ, αλλά από έναν διεθνή εγγυητή, ο οποίος να είναι σε θέση να παράσχει τη συγκεκριμένη ρευστότητα με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ιδέες υπάρχουν λοιπόν, είναι ιδέες οι οποίες πρέπει να συζητηθούν, είναι σχετικά μετρι, με, ε, εμβελίας, δεν είναι κάτι που αλλάζει σε βάθος το σύστημα, αλλά βελτιώνει ένα σύστημα το οποίο καλά δουλεύει, καλά λειτουργεί. Επανάσταση όχι, εξέλιξη ναι. Ο συνάδελφος Πόρτας και Δεν ξέρω αν ε, πρέπει να εξετάσουμε το αν υπάρχει ανάγκη για επανάσταση ή όχι. Πάντως η αδράνεια των νομισμάτων είναι ισοδυναμή με την αδράνεια των πολιτικών. Τι εννοώ. Evident. Υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στην ε, ε, σχεδόν απέραντη ικανότητα σύναψης δημοσίου χρέους στον ΗΠΑ και τις θέσεις που κατέχει το δολάριο ως, ε, στα αποθεματικά πολλών χωρών. Γι' αυτό σας μίλησα για την αδράνεια του, του ευρώ. Φαίνεται ότι το ευρώ ήδη κατέχει 20% των παγκοσμίων αποθεματικών. Παρότι δεν ε, εκδίδει ευρωομόλογα, ούτε και έχει Δημόσιο Ταμείο. αυτή η απέραντη ικανότητα σύναψης ε, χρεών που έχουν οι Αμερικανοί ε, ε, επηρεάζει όλο τον κόσμο και γι' αυτό και εγώ αναρωτιέμαι τι θα κάνουμε με την ευρωπαϊκή αδράνεια σε αυτό το τομέα. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Είπε ο συνάδελφος ότι όλοι είμαστε εδώ υπέρ της κυκλοφορίας ε, των κεφαλαίων. Εγώ θα το ομολογήσω δεν είμαι υπέρ. Αν πρέπει να αντλήσουμε ένα δίδαγμα από όλη αυτή την κρίση είναι ότι τα προβλήματα που δημιουργεί η ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων είναι ε, σαφέστατα ε, ανώτερα των πλέον εκτιμάτων που προσφέρει αυτό το σύστημα κατανομής των πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα επαναλάβω την ερώτηση που έθεσε η κυρία Περές για τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, για το φόρο αυτό επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εγώ θα κάνω την ίδια ερώτηση, αλλά τις φορολογικούς παραδείσους. Δηλαδή, ποια εμπόδια υπάρχουν τώρα όταν 80% των φορολογικών παραδείσων ε, υπάγονται στην ε, ευρωπαϊκή επικράτεια. Ποια εμπόδια λοιπόν ε, υπάρχουν, γιατί δεν υλοποιείται μια πολιτική κατάργηση των φορολογικών παραδείσων ή αλλιώς να, τα, να ε, φορολογηθούν οι εισδροές και οι εκροές κεφαλαίων ε, στις φορολογικούς παραδείσους όπως την παγκόσμια επίσημη οικονομία. Μα ποιο είναι το πρόβλημα και δεν το κάνουμε αυτό. γιατί αυτή η φορολόγηση θα έχει εθνικό χαρακτήρα, δεν θα είναι ευρωπαϊκή φορολόγηση. Οπότε δεν καταλαβαίνω ε, σε τι έγκυται ακριβώς το πρόβλημα και δεν το κάνουμε. Επίσης να κάνω και μια παρατήρηση προς τον κύριο Κλίν, τον πρόεδρο της Επιτροπής μας. Αληθεύει ότι 55% των γερμανικών εξαγωγών ε, είναι ευρωπαϊκές εισαγωγές ουσιαστικά. Ε, ε, αν όμως ταυτόχρονα <laughs> αυξηθούν και, και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών είναι το κρασί του πόρτα. Αν αυξ, αυξάνονταν λίγο και οι μισθοί, τότε σίγουρα θα κυκλοφορούσε πολύ περισσότερο το κρασί πόρτο μέσα στην Ευρώπη. Όχι, όχι, εγώ είπα 55% των εξαγωγών α, όχι είπα των εξαγωγών της Γερμανίας έρχονται από την Ευρώπη, μάλλον έρχονται από προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί από την Ευρώπη και μεταποιούνται στη συνέχεια στη Γερμανία. Θέλω να συνεχίσω με το ερώτημα που, ετέθη, που ετέθησαν από πολλούς συναδέλφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται ασφαλείς λιμένες και το δολάριο είναι το κυριότερο αποθεματικό νόμισμα. Τι θα γίνει όμως αν οι αγορές κάποια στιγμή αρχίσουν να ανησυχούν για το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών και ακολουθήσουν την γραμμή του ποπεριανού μαύρου κύκνου και έτσι βγουν από το δολάριο. Τι θα συνέβαινε στον κόσμο λοιπόν αν δούμε τον μαύρο κύκνο ενώπιόν μας. Ένα αδιανόητο γεγονός το οποίο γίνεται πραγματικότητα. Είδαμε ήδη την χρηματοοικονομική κρίση την οποία δεν μπορούσαμε να την προβλέψουμε γιατί δεν ήταν άσπρη ω κύκνο. Ήταν ένα γεγονό το οποίο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε και παρόλα αυτά συνέβη. Δεν ήταν λοιπόν λευκό κύκνο αλλά ο μαύρος κύκνος που δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, αλλά παρόλα αυτά από κάπου ενεφανιστεί. Υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο για τον ε, μαύρο κύκνο και γεγονότα τα οποία δεν προβλέπουμε συνήθως. Τι αν συνέβη κάτι τέτοιο Ιδίως αν ξέρουμε ότι το σχετικό μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας έναντι της ευρωπαϊκής οικονομίας μειώνεται σιγά σιγά στα επόμενα 10, 20, 30, 40 χρόνια. Όσο περνάει ο καιρός, εξάλλου είναι πιο πιθανό να βρούμε ένα μαύρο κύκνο. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με τα SDR, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα για ποιους λόγους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εναντίον της χρήσης των SDRs, των ειδικών τραπεζικών δικαιωμάτων και ποια είναι τα θετικά στοιχεία των δικαιωμάτων αυτών σε ένα πολυπολικό κόσμο στον οποίο ουσιαστικά είμαστε ήδη μέσα. Um, Πολλές ερωτήσεις αφορούν τις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτό το υπερβολικό πλεονέκτημα που έχουν, αν θέλετε, οι Ηνωμένε Πολιτείες με το νόμισμά τους. Όταν συζητάμε τα θέματα αυτά με εκπροσώπους της αγοράς, μας λέγουν ότι για αυτούς το δολάριο είναι ό,τι καλύτερο. Σαν παράδειγμα, αν δει κανεί τι αναπτυξιακέ ε, προοπτικέ των ΗΠΑ σε σχέση με, την, ε, με τη ζώνη ευρώ, η ΙΠΑ και φέτο και του χρόνου είναι πιο ψηλά από ότι η Ευρώπη. Αν ο κίνδυνος από τις συναλλαγματικέ ισοτιμίες στη ΣΥΠΑ δεν είναι μεγαλύτερος από ότι στην Ευρώπη ε, και δεν είναι, γιατί το πρόβλημα ίσως είναι η υπερβολική ρυθμή ανάπτυξης των αναδειωμένων χωρών. Αλλά υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι βέβαια στις χώρες αυτές και από τους ανταλλακτικούς μηχανισμούς και από πολιτικές ε, εξελίξεις μη αναμενόμενες. Και εκεί λοιπόν η καλύτερη λύση για αυτούς λένε είναι η ΙΠΑ. Και ο Σκυλακάκης λέει ότι και οι Lehman Brothers ήταν και έρχομαι τώρα στους ε, μαύρους κύκνους. Τι θα γίνει αν αλλάξει αυτό το πνεύμα των αγορών, αν θεωρήσουν οι αγορές ότι το έλλειμμα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαρκέσει. Το πρόβλημα της Καλιφόρνιας σαν παράδειγμα είναι κάτι το, ε, που δεν μπορεί να σηκώσει πλέον η οικονομία και σε άλλες πολιτείες επίσης και υπάρξει μια υποτίμηση του δολαρίου. Αυτό είναι το θέμα που έθεσα στην αρχή της πρώτης ε, παρέμβασής μου. Πρέπει να μειώσουμε τις διεθνείς ε, ελλείψεις ισορροπίας. Η οικονομία προχωρά με τέτοιο τρόπο που αν τυχόν υπάρξει μια πιθανότητα διόρθωσης, οι διορθώσεις αυτές δεν θα γίνουν με τον πιο απλό και ήμερο σε εισαγωγικά τρόπο. Αλλά πολλές φορές οι διορθώσεις μπορεί να γίνουν με καταστροφικό και απότομο τρόπο και βίαιο τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε να ληφθούν ορισμένα μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτές τις παγκόσμιες αστάθειες αν θέλετε και νομίζω ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ευρύτατη συμφωνία γύρω από αυτές τις προτάσεις. Θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός ε, προσπαθώντας να ερμηνεύσω το τι έχει στο νου της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είμαι υπεύθυνο για νομισματικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, τα σκέφτεται αυτά και έχει πει ότι δεν είναι υπέρ της επέκτασης της χρήσης των SDR γιατί θα λειτουργήσουν πληθωριστικά. Τα εκδοτικά αυτά δικαιώματα στην ουσία SDR σημαίνει τυπώνω χρήμα. Και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εγώ δεν εκφράζω την Ευρωπαϊκή Τρογγεντική Τάπεζα. Ευχαριστώ λέει ο κ. Κλίντς. Ευχαριστώ τον κύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ώρες που περάσατε εδώ μαζί μας και για όλες τις απαντήσεις που δώσατε με δεκτικό και ανοιχτό τρόπο. Στο τέλος της παρουσίασης να προσθέσω ένα πράγμα χρησιμοποιήσατε τον όρο πληθωρισμός. Είπα, ε, ακολουθούν πληθωριστικές πολιτικές για να μειώσουν ε, το επίπεδο χρέους το οποίο έχουν. Έχουν αρχίσει να τυπώνουν χρήμα. Αυτό συζητήθηκε και στη Σεούλ. Ο Γκάιτνερ είπε στους Κινέζους και το ξέρω αυτό από κάποιον που ήταν δίπλα ότι και εσείς θα πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε το επίπεδο του Γιάν Μίνμπι. Και ο Κινέζος του απάντησε ότι και εσείς θα πρέπει να σταματήσετε για κάποιες ώρες ε, τις μηχανές εκτύπωσης τις οποίες έχετε για να τραβήξετε νέο χρήμα. Λοιπόν, ανησυχώ. Ο κύριος Κλίντς λέγει ότι ανησυχεί. Ανησυχώ λοιπόν για όλες τις δυνατότητες συντονισμού που έχουμε και σε επίπεδο της ομάδας των 20 και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ζώνης ευρώ. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας κάποιες εκπλήξεις. Νομίζω ότι ε, θα περιμένουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανησυχεί για τις πληθωριστικές πολιτικές που ακολουθούνται στη ΣΥΠΑ. Για να προσθέσω σε αυτά που είπατε, σε σχέση με αυτά τα οποία κάνει το ε, Κινέζικο Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Γκάιντνερ επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα χαμηλά επιτόκια της, όπως είπανε, συμβάλλει και αυτή σε στο γενικό πρόβλημα. Αυτό το θέμα είναι αντικείμενο μιας καυτής συζήτησης μεταξύ οικονομολόγων και μέσα στη Γενική Διεύθυνση Εκφήν της Κομισιόν. Δεν έχουμε λοιπόν μια σταθμισμένη άποψη. Μπορώ να σας δώσω μόνο την προσωπική μου άποψη, αλλά αυτή δεν ανταρακλά την άποψη της Κομισιόν. Προσωπικά εγώ ανησυχώ. Ανησυχώ αλλά οι συνάδελφοί μου οι οποίοι είναι αμέριμνοι χρησιμοποιούν άλλα επιχειρήματα. Εγώ ανησυχώ γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή όταν οι άνθρωποι παρακολουθούσαν την ε, εξέλιξη των ε, συνολικών δικτών και μου λένε οι συνάδελφοί μου ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά τώρα. Τα βασικά αν αυξάνουν παραδείγματος χάρη οι νομισματικές μάζες, αυτό δεν θα οδηγήσει αδύρυτα στην ε, ανάπτυξη πληθωριστικών τάσεων. Εγώ έχω διαφορετική άποψη βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Περβόνς ε, θα ήθελε να πει το τελευταίο λόγο. Όχι ήθελα να σας ευχαριστήσω κι εγώ όπως ο πρόεδρος μα έχω πληθώρα ερωτήσεων ε, που θα μπορούσα να θέσω για ζητήματα που ούτε καν γύραμε. Παραδείγματο χάρη το θέμα της ε, δίκαιης ανταλλαγής του δίκαιου εμπορίου μάλλον εννοεί η κυρία Περές. Ε, σε σχέση με αυτά που συζητήσαμε, ε, νιώθω κάπως απογοητευμένη, αν θέλετε, και θα κλείσω με αυτή την νότα. Δηλαδή, ε, σε όλες τις αγορές έχουμε πολύ ρευστότητα που ρίξαμε στις αγορές μετά την κρίση, αλλά ε, ελοχεύει ένα κίνδυνο να δημιουργηθεί μια υπερμεγέθη κερδοσκοπική φούσκα, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώ πού πήγανε τα λεφτά αυτά, πού πήγε αυτή η ρευστότητα. Στα πλαίσια του G20, Γίνεται μια συζήτηση που όμως δεν οδηγεί ποτέ σε συμπεράσματα. για να βρεθούμε στην ε, κρίση στην οποία βρεθήκαμε. Υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες, ε, δεν υπάρχουν μονοριακά προβλήματα. Ε, φοβούμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε την κρίση ώστε να επαναπροσανατολίσουμε τη λειτουργία των αγορών και να εξυπηρετούνται μακροπρόθεσμα πλέον τα συμφέροντά μας. Διότι εντάξει, συζητάμε για το ρεμίμπι και τη σχέση του με το δολάριο, ωραία. Αλλά τι κάνουν οι μεν και οι δε ούτω ώστε οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ να εξυπηρετούν τι πραγματικέ ανάγκε τη πραγματική οικονομία που είναι τεράστιε. σω το δείπνο να, συζητείτε, να συζητούνται τέτοιου είδου θέματα, αλλά δεν αλλάζει και τίποτα. Η βασική παίκτε των χρηματοπιστωτικών αγορών συνεχίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τελευταία παρατήρηση για τη λειτουργία των ε, υποδομών. Παρότι υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο μέσα στην έκθεση, δεν το συζητήσαμε καθόλου. Το ερώτημα είναι αν επιθυμούμε παγκόσμια διακυβέρνηση και σε ποιο επίπεδο. Ε, φτάνει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ή δεν επαρκεί. Αν ε, είναι να υπάρξει παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να ε, την αναλάβουν και να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο διακυβέρνηση, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στην ε, χρηματοπιστωτική διάσταση, γιατί αλλιώ δεν θα λάβουμε υπόψη ε, άλλες εξίσου σημαντικές συνιστώσεις. Αν ασχοληθούμε τέλος πάντων μόνο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ομάδα G20 θα έπρεπε ή θα μπορούσε να ε, αναδειχθεί σε εκτελεστική επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί δείτε πώς λειτουργεί, δείτε ε, ποιος, ε, ποιος διοικεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομίζω ότι δεν θα βγάζαμε άκρη με την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση αν οι παίκτες που βλέπουμε τώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λάμβαναν αυτό το ρόλο. Φαίνεται να να επιχειρώνεται αυτά τα οποία είπα εγώ και την ανησυχία μου ότι όλα αυτά έχουν προσθεθεί στο σύστημα και επομένως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο διεξόδου. Κάτι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν όλα, όλες αυτές οι νέες παράμετρε στο σύστημα. Μου λένε οι συνάδελφοί μου ότι ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους, ότι η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού τομέα και η μεταρρύθμιση έχει αλλάξει τη δομή του συστήματος. Ελπίζω να έχουν δίκιο και να μην αναπτυχθούν πληθωριστικές πιέσεις σε λίγα χρόνια. Γιατί όπως ξέρετε στο παλαιομοδίτικο σύστημα στο οποίο εγώ γνώριζα η στέρηση μέχρι να αναπτυχθούν πληθωριστικές πιέσεις ήταν 2-3 χρόνια. Απλώς για να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα και σας λέω και πάλι αυτά είναι τελείω προσωπική μου άποψη. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει και ο πρόεδρος.